Good morning. Καλημέρα σε όλους, αλλά και σε όλες. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ειδική ακρόαση για την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά από αυτήν κυρίες και κύριοι βουλευτέ που συμμετέχετε στο σεμινάριο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαιτέρως τις προσωπικότητες οι οποίες ε, έχουν ε, έρθει και κάθεται εδώ στο βήμα δίπλα μου και δει την Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα την κυρία Βίβια Ρέντινγκ, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος ε, μιας ε, ομάδας εργασίας, μιας συνεδρίας εργασίας ουσιαστικά που γίνεται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την Επιτροπή των Θεμελιωδών ε, Ελευθεριών, μάλλον πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Χθες ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα και επικοδομητικά για το ρόλο του χάρτη ως ένα σημείο αναφοράς για το μελλοντικό νομοθετικό έργο που ως ε, τακτικοί νομοθέτες ε, έχουμε ως ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ιδίως σε έναν τόσο σημαντικό τομέα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως είναι η προστασία του θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από την δικαστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το δικαστήριο, αλλά όχι μόνο και από τις ε, δικαστικές εξουσίες ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόν τον διαδραστικό και αμοιβαίο διάλογο που είναι πάρα πολύ εμπλουτιστικό, στον οποίο έχουν ε, τα διάφορα δικαστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους, στο πλαίσιο των νομών κύκλων για την προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύουν τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την έννοια ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τρίτη συνεδρία σήμερα αφορά τον χώρο ελευθερία δικαιοσύνη και ασφάλεια και θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε ό,τι αφορά επίσης ε, την κοινωνική ε, και πολιτική προστασία, τις ε, διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσοι βουλευτές συμμετέχοντες θέλετε να λάβετε το λόγο, σας ενημερώνω ότι θα πρέπει απλά να ενημερώσετε το Προεδρείο. Κάντε ένα σήμα, σηκώστε το χέρι, στείλτε μας ένα σημείωμα αναφέροντας το όνομά σας και την οργάνωση, το φορέα που εκπροσωπείτε σε αυτό το σεμινάριο σε αυτή την ακρόαση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στην Επίτροπο Vivian Ρέντινγκ και αμέσως μετά θα έχουμε έναν γύρο ερωτήσεων τις οποίες θα απαντήσει η Επίτροπος. Κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη θέση ενισχύει της συνθήκης Λισαβόνας καταφέραμε, πετύχαμε μία ιστορική αλλαγή, διότι τώρα έχουμε ένα, μια δεσμευτική χάρτα που είναι η απαρίθμηση που έχουμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα όμως πρέπει να την εφαρμόσουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο η Κομισιόν μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα κάνει μια δήλωση όπου θα περιγράφει τη στρατηγική της για την εφαρμογή της χάρτας. Ο κύριος στόχος εδώ είναι να, την καταστήσουμε, να όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα που αναφέρονται στη χάρτα για όλους όσους ζουν και διαβιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη της Ένωσης, η συνυπογραφή από την Ένωση στην, ε, στην ε, Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο πρόκειται επίσης σύντομα να γίνει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν παρεμβαίνει σε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφόσον η Ένωση είναι υποδειγματική στην εφαρμογή το, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Άρα η χάρτα θα είναι ο μπούσουλας των πολιτικών αυτών και της εφαρμογής των μέσα στο συλλογικό σώμα της Κομισιόν πρέπει η χάρτα να καθοδηγεί την δράση όλων των υπηρεσιών. Ίσως να θυμάστε ότι στις 3 Μαΐου όλοι οι επίτροποι υποσχέθηκαν επίσημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ορκίστηκαν μάλιστα, να σεβαστούν την χάρτα κατά την εφαρμογή των καθηκόντων τους. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Θέματα ασφαλείας εδώ πρέπει να δείξουμε τη δέσμευσή μας προς την χάρτα στην πράξη. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να συμβαδίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όσο ισχυρότερες είναι οι εγγυήσεις που θα δίνει η Ένωση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο περισσότερες θα είναι οι ευκαιρίες της Ένωσης να προοδεύσει, να πετύχει πρόοδο πράγματι στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τορομοκρατίας. Αυτό μάλιστα γράφεται ρητά από το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Οι αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες πρέπει να γίνονται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό. Πρώτη μου προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ένωση όταν νομοθετεί θα λαμβάνει πάντοτε υπόψη της ως προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την αρχή ήδη της διαδικασίας, όταν δηλαδή η Κομισιόν προετοιμάζει μια πρόταση. Η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να επιτηρεί την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελπίζουμε ότι έτσι το σύνολο της Κομισιόν θα πετύχει την εφαρμογή ενός γενικού κλίματος σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδείγματος χάρη, οι πράσινες βίβλοι της Κομισιόν πρέπει πάντοτε να σέβονται τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι έτσι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το κίνητρο και εκείνοι να το πράξουν. Και έπειτα έρχεται η επόμενη φάση, η αξιολόγηση της εφαρμογής των, της νομοθεσίας στο θέμα ακριβώ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ενδυναμωθεί η διάσταση αυτής της αξιολογικές μελέτες που πρέπει να ταυτίζουν ποια θεμελιώδη δικαιώματα αφορώνται και πώς γίνονται σεβαστά. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει επίσης να περιγράφουν σε τι βαθμό υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων και τι πρέπει να γίνει σε τέτοια περίπτωση. Και λέγοντας αυτό εννοώ ότι αυτό δεν θα περιορίζεται στην Κομισιόν. Πρέπει και το Συμβούλιο να κάνει τα ίδια. Παραδείγματο χάρη σε θέματα ποινικού δικαίου όταν θέλει να προτείνει κάτι το Συμβούλιο. Συνήθως δεν γίνονται αξιολογήσεις κανενός είδους μέχρι τώρα. Νομίζω όμως ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει να γίνεται και για αυτά τα θέματα μία τακτική και κανονική για τη γενική επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και μία δεύτερη χωριστή ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η αντίληψη της χάρτας ως μπούσουλα είναι κάτι που πρέπει να αφορά ολόκληρη την νομοθετική διαδικασία ώστε το τελικό κείμενο, το νομοθέτημα δηλαδή, μετά από τη συζήτηση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου επίσης να συμβαδίζει με την χάρτα. Και εδώ έρχεται το θέμα της συλλογική ευθύνης όλων των θεσμικών οργάνων. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι οποιοδήποτε τελική συμβιβασμή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμβαδίζουν και με τη χάρτα. Αυτό επίσης το έχει το Συμβούλιο στη δήλωση ή στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πρέπει λοιπόν σε διαθεσμικό επίπεδο να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο ή τι αλλαγές, τι τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν, πώς θα αξιολογούμε τις τροπολογίες και τους συμβιβασμούς χωρίς να αγνοούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσουν και την εμπειρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Δημοσίων Ελευθεριών. Και αυτό θα ισχύει και για τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Παραδείγματος χάρη στα θέματα της δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και για την αστυνομική συνεργασία. αν και ελπίζουμε να μην χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες, όταν χρειάζονται θα πρέπει να εξετάζεται και η διάσταση του σεβασμού του χάρτας των θεμελιωδών. Έχουμε λοιπόν το κείμενο, το έχουν ψηφίσει τα όργανα και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί, να μεταφραστεί σε ενωσιακή νομοθεσία και να μεταφερθεί στην εθνική. Και γι' αυτό η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με τις συνθήκες για να διασφαλίσει το σεβασμό της χάρτας και από την εθνική νομοθεσία που θα μεταφέρει την ενωσιακή. Σας έχω ήδη πει εδώ ότι δεν θα διστάσω να αρχίσω προσφυγές για παράβαση και παράληψη εάν σημειωθούν παρατυπίες. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή σας συνεδρίαση της ακρόασης με συμμετοχή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Ακαδημαϊκού Κόσμου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να τονιστεί η ανάγκη για περισσότερη και ακριβέστερη πληροφόρηση. Η υπηρεσία αυτή εδώ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο δίνοντάς μας συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση και στις 27 χώρες μέλη στα θέματα που έχει δικαιοδοσία βέβαια η Ένωση. Οι εμπειρογνώμονες από την κοινωνία των πολιτών έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από εμά επιτόπου και χρειαζόμαστε και τη δική τους συμβολή. Για να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες βέβαια η Κομισιόν θα δημοσιεύει ετησίως μια έκθεση για την εφαρμογή της χάρτας. Ιδιαίτερα βεβαίως από εκ μέρου των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Θα παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή της σε τομείς όπου έχει δικαιοδοσία η Ένωση. Πρέπει πάντοτε να το προσθέτω αυτό. Και θα αναφέρει και παραδείγματα της εφαρμογής της χάρτας ε, σε συγκεκριμένους τομείς της δράσης της Ένωσης. Αυτή η ετήσια έκθεση βέβαια θα επιτρέπει και μία ετήσια συζήτηση για σχεδιασμό και πολι... της πολιτικής στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τι ελλείψεις μπορεί να υπάρχουν κλπ. Θα έχετε καταλάβει λοιπόν από όλα αυτά ότι Αυτό δεν αφορά μόνο τον αρμόδιο ή την αρμόδια επίτροπο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι θέμα που αφορά όλα τα θεσμικά όργανα και όλους και όλες τους ενδιαφερομένους και ενδιαφερόμενες. Πρέπει η χάρτα να εφαρμοστεί στην πράξη διότι δεν είναι μόνο ένα θεσμικό μια θεσμική οντότης αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες μέλη και όλα τα θεσμικά όργανα. Επειδή είναι νομικά δεσμευτική, αποτελεί και την απαρχή μιας νέας φάσης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και είμαι βέβαιη ότι μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου, των χωρών μελών και του Συνοβουλίου για να δημιουργηθεί επιτέλους ένα ολόκληρο κλίμα, μια κουλτούρα κουλτούρα θεμελιωδών δικαιωμάτων για να το πω έτσι. Και μάλιστα καθημερινή. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ. Θα κάνουμε συζήτηση τώρα. Η και πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι η συγγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής ΛΥΜΕ για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ε, ακρόαση αυτή και χτες ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά και σήμερα ευχαριστούμε την Επίτροπο που κατάφερε να έρθει μαζί μας παρόλο που δεν είναι και ιδιαίτερα καλά σήμερα Συμφωνώ απόλυτα με, το, με αυτά που είπατε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πραγματική ουσιώδη εφαρμογή της χάρτας. Έχουμε τώρα ένα έγγραφο νομικά δεσμευτικό, πολύ σύγχρονο. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτή η διήμερη ακρόαση εδώ και η έκθεσή μου πράγματι προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το ρόλο που θα παίζει στο μέλλον η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να διευκρινίσουν και κάποια πρακτικά πράγματα, ποιος θεσμός θα κάνει τι, ποιο θεσμικό όργανο και τι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τα θεσμικά όργανα, δημιουργήσαμε τους μηχανισμούς, τώρα πρέπει να μπούμε και σε λεπτομέρειες. Χάρηκα που είπατε ότι θα υπάρχει μηδενική ανοχή για τις παρατυπίες και τις παραβάσεις και ο ρόλος της Κομισιόν είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή και να κυρώνει ε, παρατυπίες και τα λοιπά. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν ε, και τα επαρκή στοιχεία για να παρθεί τελική απόφαση. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τώρα γιατί είναι σημαντικό για την έκθεσή μας εδώ στο Κοινοβούλιο πω τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει και τι θα συμβεί ακριβώς αν διαπιστωθεί αν θέλετε παρατυπία πρόεδρος αν, ε, κυρία Επίτροπε ας, πάρω, ακούσουμε μια-δυο ακόμη ερωτήσεις και μετά απαντάτε συνολικά η κυρία Αντζολίλη Ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Ρέντινγκ. Χαιρόμαστε ε, θυμίζω παλιότερα που είχαμε πάρει την απόφαση για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τότε είχε γίνει σχετική πρόταση από την Κομισιόν ε, χαρήκαμε για την πρόταση αυτή αναγνωρίσαμε την αξία της και για πολλά χρόνια λέγαμε ότι περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ και η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και η χάρτα των ε, θυμαλαιοδών δικαιωμάτων γιατί θεωρούσαμε ότι με την χάρτα αυτή θα συμπληρωνόταν μια Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή νομική βάση αν θέλετε για να προστατεύσουμε πλήρως τις ε, ε, μειονότητες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα αναφερθώ σε πολλά πράγματα που ίσως ακόμη πρέπει να συζητηθούν. Απλώς θα ήθελα να ρωτήσω τι πιστεύετε, πώς πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί θα επηρεαστεί η προστασία των εθνικών μειονοτήτων από τη χάρτα αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο που βρίσκεται μαζί μας εδώ σήμερα. Και επειδή τη γνωρίζουμε την κυρία Επίτροπο, ε, έχουμε, έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και θα μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά η χάρτα σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τι... Ε, βεβαίως υπάρχουν βεβαίως έχουμε τις νομικές βάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να ε, βασιστούμε σήμερα αλλά θα θέλαμε να δούμε και στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών πως θα ε, βιώσει κανείς την εφαρμογή της χάρτας. Κύριε Επίτροπε Πώς λογαριάζετε να ελοποιήσετε πρακτικά τη χάρτα αυτή, πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει με ποιους τρόπους για να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες από α, παρατυπίες και παραβιάσεις. Γιατί η δικαστική οδό σε πάρα πολλές χώρες είναι μακρόχρονη και επίπονη. Κυρία Μπότσκολ, ευχαριστώ να πω καταρχάς ε, ότι είναι πάρα πολύ ε, καλό που βλέπουμε εδώ την Επίτροπο που προσωπείται και που ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσία της. Να κάνω κάποιο σχόλιο. Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις μελέτες επιπτώσεων και τις αξιολογήσεις. Καλό θα ήταν όμως να περάσουμε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε κατά πόσον τα προβλεπόμενα μέτρα είναι ή δεν είναι αντιφατικά σε σχέση με αυτή τη χάρτα. Θα ήθελα επίσης να δω πώς όλα αυτά θα τα ε, υλοποιήσουμε ενεργά. Πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση θα πρέπει να δούμε τι αντιφάσεις υπάρχουν για το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται είναι οι προτάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται ε, στα ίσα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεν φάνηκε ιδιαίτερα θετικό το Συμβούλιο. Έδειξε κάποια συντισταγμούς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φορεί εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω το Συμβούλιο τη Ευρώπη, παραδείγματο χάρη, που ασχολούνται με τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει σχέση με τέτοιου φορεί και τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθε, α πούμε, στην Εξεταστική Επιτροπή είδα, μάλλον είδα ότι ξεκίνησε μια Εξεταστική Επιτροπή κατά σεξουαλικών ε, κακοποιήσεων παιδιών. Ε, τι μπορεί να κάνει, έχει πρόθεση να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι σημαντικό και για του πολίτε και για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο, κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται μαζί μας εδώ η Επίτροπος Ρέντινγκ. Θα ήθελα να ε, της υποβάλω ένα συγκεκριμένο ερώτημα γιατί και η κυρία Ρέντινγκ ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Η σημερινή κατάσταση που βιώνουμε στην Ευρώπη απαιτεί η νέα χάρτα πράγματι να χρησιμοποιηθεί και σε όλες τις νομοθετικές ε, δράσεις των κρατών μελών. Ρωτώ λοιπόν, η υφιστάμενη οδηγία η οποία την οποία έχουμε και η οποία απαγορεύει διακρίσεις βάσει εθνοτικών χαρακτηριστικών ε, μιλά για, για αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά δεν μιλά για γλωσσικές διαφορές λοιπόν η χάρτα θα βελτιώσει την κατάσταση αυτή δηλαδή από εδώ και μπρος όταν θα ε, εφαρμόζουμε την οδηγία κατά των διακρίσεων σε κάποιο κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη γλωσσική προέλευση ή όχι. Yes, please. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαρίσες Το πρώτο άρθρο της χάρτας υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να τη χάνει σεβασμού και προστασίας. Όσοι όμως ζουν σε μεγάλη τεράστια ακραία ανέχεια ε, δεν την χάνουν του σεβασμού αυτού. Τα οικονομικά, πολιτιστικά αλλά και πολιτικά τους δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Πρόκειται λοιπόν για σοβαρή παραβίαση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ερωτώ λοιπόν κυρία Επίτροπε, η Κομισιόν προτίθεται να κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση αυτής της ακραίας ανέχειας ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρω ότι η Υπηρεσία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θέλει να κάνει κάτι για να αναπτυχθεί, να δημιουργηθεί αυτό που είπατε στο τέλος, μια ολόκληρη κουλτούρα δικαιωμάτων. Ε, αυτή νομίζω πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την καταπολέμηση της ακραίας ανέχειας ως πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Επίτροπος. Ε. Η κυρία Κάλ ρώτησε για το κατά πόσον και πότε θα δημοσιοποιηθούν οι εκθέσεις. Μπορώ να σας πω κυρία Κάλ πολύ συγκεκριμένα ως απάντηση στο ερώτημά σας ότι θα έχουμε δύο εκθέσεις. Η πρώτη θα είναι μια ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρεται η πολιτική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς επίσης και η υλοποίηση των πολιτικών αυτών από πρακτικής πλευράς στα κράτη-μέλη. Άρα, το πιο θεωρητικό κομμάτι ε, του πώς δηλαδή θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και μετά θα έχουμε μια ετήσια έκθεση πολύ πιο συγκεκριμένη ετήσια, όπως είπα, έκθεση, στην οποία θα εξετάζεται το πώς εφαρμόζεται πρακτικά η πολιτική αυτή. Λειτουργεί, έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει. Πού χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις. Πού μπορούμε να πούμε ότι ορίστε να ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να το ακολουθήσουμε και το καθεξής. Επομένως η υλοποίηση της χάρτας από πρακτική πλευρά. Η ανακοίνωση θα είναι άπαξ. Ενώ η αιτήσια έκθεση θα γίνεται κάθε χρόνο, θα εκπονείται κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά θα δημοσιοποιηθούν από κοινού η ανακοίνωση με την ετήσια έκθεση. Δηλαδή το σημαντικό, η σημαντική δημοσίευση φέτος θα είναι αυτή της ανακοίνωσης γιατί υπάρχει μια μικρή περίοδος ανάλυσης. Η έκθεση η ετήσια του 2011 θα είναι η σημαντική ετήσια έκθεση, όχι αυτή του 2010. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα ε, γίνει η δημοσίευση δηλαδή ε, τέλη Οκτωβρίου, το φθινόπωρο πάντως. Όταν έχω, κυρία Ισηγήτρια, τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα σας ενημερώσω σχετικά για να προετοιμαστείτε κι εσείς, να προετοιμάσετε το έργο σας για την κυρία Αντζελίλη για τα δικαιώματα των μειονοτήτων προβλέπεται στο άρθρο 2 της ε, συνθήκης προστασία των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων αλλά και στο άρθρο 21 της χάρτας. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά ως προς τον τομέα αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή πλέον ε, έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου εδώ και κάποιους μήνες, έχω λάβει περίπου 600 ερωτήσεις, έτσι καταλαβαίνετε περί τενός πρόκειται. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μου το μόνο που κάνουν είναι να απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, έχω υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο ότι θα υπάρξει μια λεγόμενη μονοαπευθυντική θηρίδα, ένα one-stop shop στη νέα γενική διεύθυνση η οποία θα συγκροτηθεί την 1η Ιουλίου. Το Κοινοβούλιο θα έχει λοιπόν αυτή την μόνο του θηρίδα για τα ζητήματα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων από την, τον Ιούλιο και μετά. Για το επόμενο στάνσε, πώς επηρεάζουμε και πώς ελέγχουμε. την εφαρμογή των, και την υλοποίηση των δικαιωμάτων σε επίπεδο κρατών μελών. Φυσικά, γι' αυτό χρειαζόμαστε ανάλυση, ανάλυση της κατάστασης στα κράτη-μέλη, του τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Αυτό θα το συμπεριλάβουμε μετά στην ετήσια έκθεση. Το πώς εμείς τώρα, τα θεσμικά όργανα, εφαρμόζουμε τη χάρτα, αλλά και πώς το Συμβούλιο, πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τη χάρτα. Αν καταστεί απαραίτητο και αν δεν καταφέρνουμε να λύσουμε, να λύσουμε αλλιώς το πρόβλημα, θα κινήσουμε διαδικασία επί παραβάση. Σε ό,τι αφορά την κυρία που μίλησε για τις μελέτες επιπτώσεων, αξιολόγηση των επιπτώσεων, έναν κανόνα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οποιαδήποτε πρόταση νομοθετικού περιεχομένου υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλεται πρώτα σε αξιολόγηση των επιπτώσεων, η οποία δεν είναι μόνο σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής επίπτωσης που θα έχει το συγκεκριμένο νομοθέτημα αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο κριτήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά το φθινόπωρο, στα κείμενα που θα σας παρουσιάσω, θέλουμε να υπάρχει και αυτό το κομμάτι της αξιολόγησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να αποτελεί ένα κανονικό κομμάτι της νομοθεσίας της ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο πρέπει να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια νέα συνθήκη και υπάρχει ο χάρτης πια. Πρέπει να τους το επαναλαμβάνουμε σε τακτά διαστήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Σύμβουλιο της Ευρώπης, γνωρίζεται ότι έχω την εντολή να διαπραγματευθώ την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης ε, με τακτικά με το Συμβούλιο της Ευρώπης για το θέμα αυτό, την κυρία Μπάουερ, η οποία μίλησε για το ζήτημα των γλωσσών πολύ σωστά, όπως λέτε, δεν συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες κατά, για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ωστόσο, αναφέρεται στο άρθρο 21 της χάρτας που απαγορεύει ρητός οποιαδήποτε διάκριση λόγω γλώσσας ε, ή ε, ανήκει σε μια συγκεκριμένη μειωτική ομάδα. Ο χάρτης τώρα αυτός έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα εφαρμόζεται, θα εφαρμοστεί. Ωστόσο τα κράτη-μέλη παραμένουν ε, υπεύθυνα σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για την εσωτερική τους πολιτική σε θέμα γλωσσών συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ημενοτικών γλωσσών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κοινοτική νομοθεσία που να ρυθμίζει τη χρήση των γλωσσών. Η Επιτροπή θα παρεμβαίνει όποτε προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Και θα ήθελα στο θέμα των γλωσσών να υπενθυμίσω τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφυρακών και Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και τη Σύμφαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, φτώχειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναλύει διεξοδικά όπως έχει πράξει το πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και γνωρίζω ότι ο κύριος Άντορ, ο αρμόδιος επίτροπος για τα κοινωνικά θέματα, εκπονεί επί του παρόντος μια στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας ανέχειας, μεταξύ άλλων. Αυτό θα είναι και μια συγκεκριμένη πράξη στο πλαίσιο της στρατηγικής μια συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Ο Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ακούσαμε ότι δεν είστε πολύ καλά σήμερα. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχόμαστε περαστικά. Και προχωρούμε. Σας αποχαιρετούμε και χαιρετούμε τον επόμενο μιλητή. Now let's, let's according to the agenda by giving the floor to Mr. ακολουθούμε λοιπόν την ε, ημερήσια διάταξη και δίνουμε το λόγο στον κύριο Τζέραμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε κυρία Ρέντινγκ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να έρθω σήμερα εδώ στην ακρόαση αυτή η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη διότι ακόμη βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας και της εφαρμογής της. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε το ρόλο της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανάγκη εφαρμογής του. το να τηρηθεί απόλυτα η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι μεγάλη πρόκληση κυρίες και κύριοι. Στο Ευρωβαρόμετρο είδαμε πρόσφατα ότι 62% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το πιο σημαντικό, την πιο σημαντική αξία που πρέπει να προστατεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να πω μερικά πράγματα για το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τη χάρτα να δουλέψει σωστά. Πρώτα-πρώτα, τα δικαιώματα που βρίσκονται στα χαρτιά μας πρέπει να γίνουν πραγματικά δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να είναι περήφανη για τη χάρτα αυτή η οποία είναι απλή, σαφής, κατανοητή και ουσιαστικά δίνει στους Ευρωπαίους ένα ε, Bill of Rights όπως θα λέγαμε στα αγγλικά ε, μία βάση πάνω στην οποία να μπορούν να, ή να πρέπει να βασιστούν όλες οι μελλοντικέ νομοθετικές δράσεις όλων των κρατών μελών Είπα, αναφέρονται λοιπόν όλα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στη χάρτα αυτή και ένα τα δικαιώματα αυτά είναι η να πρεπει να βασιστουν ολες οι μελλοντικε νομοθετικες δρασεις ολων των κρατων μελων αναφερονται λοιπον ολα τα βασικα ανθρωπινα δικαιωματα στη χαρτα αυτη και ενα τα δικαιωματα αυτα ειναι η ιδιωτικοτητα της το δικαίωμα για ιδιωτική ζωή. Και αυτό είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να το επιβάλλουμε. Υπάρχουν τέτοιου είδου δικαιώματα λοιπόν, τα οποία κάπου μέχρι τώρα ήταν απλώ φιλοδοξίε και ωραία λόγια χωρίς να εφαρμόζονται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι τα δικαιώματα που υπάρχουν στα διάφορα χαρτιά τώρα θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Η μη, το να μην υπάρχουν διακρίσει. Βεβαίω υπάρχουν οι οδηγίε για την ε, τα πολέμηση των διακρίσεων. Αλλά εδώ μπορούμε να πάμε ακόμη πιο πέρα. Ανησυχούμε για το γεγονός ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Δεν γνωρίζουν την, το πώς να προστατευθούν ή το τι υπάρχει σαν δικαίωμα για να προστατευθούν από τις διακρίσεις. Η, βρήκαμε από ε, πρόσφατα στοιχεία ότι μόνο 25% των πολιτών γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και την ανάγκη να προστατεύονται από διακριτική μεταχείριση λόγω φιλετικής προέλευσης, λουσικής προέλευσης όπως έλεγε προηγουμένως κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα γνώσεων και έτσι 82% των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης τα τελευταίους 12 μήνες δεν ε, προσέφυγαν σε κανένα φορέα ή αρμόδια αρχή που θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Κάτι το αντίστοιχο σχετίζεται και με την... Ε, ε, κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και για, να λέγεται και στην έκθεση για την ομοφιλοφιλία που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Και το μίσος για τους ομοφυλόφιλους που φαίνεται να υπάρχει. Η, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ατιμορρησία των δραστών και μη προστασία των θυμάτων. Άρα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα εδώ. Πρώτα πρώτα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε κάποιους φορείς που μπορούν να τους προστατεύσουν, μπορούν να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη και κυρίως πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους, τους πιο περιθωριοποιημένους, να τους εξηγήσουμε τι μπορούν να κάνουν αν δεν γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Όλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, οι κυβερνήσεις, οι φορείς ε, της ε, η κοινωνία των πολιτών, Όλοι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά στο κέντρο βρίσκεται πάντα ο πολίτης. Και πρέπει να επικοινωνήσουμε λοιπόν με τους πολίτες και να τους πούμε ακριβώς πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν, να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό λέγεται και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Δεύτερο θέμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να είναι στο κέντρο και στη βάση όλων των νομοθετικών ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όλες τις αναλήψεις νομοθετικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, για και ε, για οτιδήποτε θέμα και θα ήθελα να τονίσω εδώ τη συνθήκη για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες για των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ε, αναπηρίες η αντιπρόεδρος Ρέντινγκ ανέφερε πολλά ε, σημεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάρα πολύ ε, σοβαρά στη μελλοντική νομοθετική δουλειά της Ένωσης και στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου από την αρχή ήδη για να μπορούν να ενταχθούν και όλες τις νομοθετικές προσπάθειες. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα κράτη-μέλη και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τον έλεγχο της ε, συμμόρφωσης όλων προς την ε, χάρτα αυτή. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης λέγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιείται και η υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και η προσφυγή στην, στην υπηρεσία αυτή. Πράγματι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί αυτή τη στιγμή και μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να κάνει αναλύσεις για τα στοιχεία, αξιολόγηση της δράσης στα διάφορα κράτη-μέλη, μπορεί να βοηθήσει στην εκπόνηση πραγματικών νομοθετικών πράξεων που σέβονται ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τρίτο θέμα που ήθελα να τονίσω είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να συμμετάσχουμε στην εφαρμογή της χάρτας. η εφαρμογή της χάρτας δεν είναι ένα project ευρωπαϊκό. Είναι κάτι όπου όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι πολίτες, όλα τα σχολεία, όλοι οι επιθεωρητές των σχολείων, ο καθένας θα πρέπει να συμμετάσχει. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και σε εθνικό επίπεδο προφανώς ε, θα πρέπει να γίνουν τεράστιες προσπάθειες και εδώ ακριβώ βρίσκεται η πρόκληση το 2009 16.000 αιτήσει κατετέθησαν στα 27 κράτη-μέλη ε, ε, για ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, προσφυγές, ε, 16.000 ε, προσφυγές έγιναν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσέφυγαν στο Στρασβούργο για να προστατευθούν. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς. Υπάρχουν εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν άλλες οργανώσεις οι οποίες θα έπρεπε να εμπλακούν και οι οποίες ίσως έχουν κάποιες ελλείψεις σε προσωπικό ή άλλους πόρους ε, οι οποίες θα πρέπει τις οποίες επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά κοινοβούλια, ναι. των οποίων ο ρόλο ενισχύεται στη συνθήκη της Λισαβόνα. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το, τα θεμελιώδη δικαιώματα θα έπρεπε να μπαίνουν κάθε φορά στην ημερήσια διάταξη των κοινών συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εκεί θα μπορούσαν να εμπλακούν και οι εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίω, διατρέχουμε μια σοβαρή οικονομική κρίση και γι' αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο να παρεμποδιστεί κάπως ο ρόλος των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υποστηρίζονται οικονομικά οι βασικοί φορείς που προστατεύουν τα σεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και να μην ξεχνάμε και το τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Έχουν αρμοδιότητα σε τομείς που επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητα των πολιτών να συνειδητοποιήσουν και να απαιτήσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει και αυτή να συμμετάσχει στην εφαρμογή της χάρτας. Και ε, εκεί θα πρέπει να βοηθήσει και η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσπαθεί να προωθήσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλοι αυτοί οι φορείς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην υπόθεσή μας για να διασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό και να ε, κάνουν πραγματικά κοινό στόχο την προστασία των σεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν συμπεράσματι χαιρετίζουμε τη χάρτα των σεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς αλλά δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει να αγωνιστούμε για να δώσουμε ζωή στο καινούριο αυτό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζω με την ομιλία μου αυτή να σας έδωσα μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ομιλητή, στον κύριο Τζαν Τζαράμ από την είπα τη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και στον κύριο Ροντοτά ο οποίος ήταν μέλος της συνέλευσης που ε, πόνισε, που συνέταξε τη χάρτα των σεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο κύριος Τζάραμπ, λοιπόν, πρώτα-πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την ευγενή πρόσκλησή της προς την υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην σημερινή συνεδρίαση που συζητάει για το ρόλο της Χάρτας Θεμελιωδών και στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας Δικαιοσύνης με την ε, έγκριση της χάρτας αυτής καθώς και της, Ευρωπαϊκής, της δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση έχει βελτιωθεί ήδη και μάλιστα τρομερά. Η ε, θέση ενισχύει της συνθήκης Λισαβόνας που καθιστά τη χάρτα νομικά δεσμευτική για τα κράτη-μέλη είναι απτή απόδειξη της θέλησης της Ένωσης να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ελευθερίες που προβλέπει. Τα δικαιώματα της χάρτας συμπεριλαμβάνουν και την υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη να τα τηρούν και τα περισσότερα από αυτά τα εμπνεύστηκαν οι συντάκτες τους από υπάρχοντα έγγραφα όργανα και οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά με διευρυμένη έννοια όπως ας πούμε την ειδική προστασία που πρέπει να χορηγείται σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες. Η χάρτα όμως έχει περιορι... Ε, περιορίζει τη δράση της στις χώρες της Ένωσης και στα θεσμικά της όργανα. Οι διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν συνυπογράψει οι χώρες μέλη δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς και όπως είπε και ο κύριος Σέρμ και η ίδια η Ένωση πρόσφατα συνυπέγραψε την πιο πρόσφατη διεθνή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σύμβαση για τους αναπήρους. Τα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνει η χάρτα καθώς και άλλες διεθνείς συμβάσεις που συνυπόγραφουν τα κράτη-μέλη είναι συμπληρωματικά. Η χάρτα θα είναι στο μέλλον ε, η πηξίδα ή ο μπούσουλας για τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται γενικότερα και για τις διεθνείς υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Άρα και για τα θέματα του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφαλείας. τα διεθνή σώματα επιτήρησης των προβλεπομένων από διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελέσουν την έμπνευση και για την επιτήρηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αξιολόγησή τους εθνικά. Έχω λοιπόν την τιμή και την ειδονή να είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω ότι φέτος στην ετήσια συνεδρίαση των προέδρων αυτών των σωμάτων επιτήρησης για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία εκτός Γενέβης εδώ στις Βρυξέλλες 1η και 2 Ιουλίου θα οργανωθούν δύο δημόσιες ακροάσεις με εκπροσώπους και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών. πρέπει να τονίσω ότι θα αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα από τις επισκέψεις των επιτηρητών στις χώρες. Θα έχουν το δικαίωμα αυτές να δηλώσουν τι προόδους έχουν σημειώσει και τι ελλείψεις έχουν παρατηρήσει. Μετά από αυτή την αναθεώρηση γίνονται κάθε φορά και συστάσεις προς τις χώρες μέλη που θα αφορούν κυρίως τα θέματα που θέτει και η χάρτα. Και αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο για να υπάρχει συνέπεια και συνοχή στην πολιτική, στη διεθνή πολιτική ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επιτήρηση που προβλέπει η Ένωση για την εφαρμογή της ίδιας της, της χάρτας είναι κάτι το πολύ σημαντικό των δικαιωμάτων που αναφέρει η χάρτα αλλά και τα διεθνή πρότυπα. Μια τέτοια επιτήρηση εάν γίνει όπως πρέπει θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και επί της δέσμευσης της Ένωσης για την προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτός αυτής. Και έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Διότι αν η Ένωση δεν επιτηρήσει πρώτα τα ίδια της τα κράτη-μέλη και δεν τονίσει τις ελλείψεις τους, ενώ θα πράξει το ίδιο διεθνώς, αυτό θα σημαίνει ότι θα μειώσει την αξιοπιστία της, θα κατηγορηθεί για διαφορετικά μέτρα και σταθμά και θα καραδαρακωθεί διεθνώς. Το γενικότερη αυτή έννοια λοιπόν του χώρου ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης είναι κάτι που αφορά και την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση ας πούμε τα δικαιώματα των μεταναστών, άσυλο, προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξισορρόπηση μεταξύ ασφαλείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την καταπολέμηση της τυρομοκρατίας και φυσικά και θέματα που αφορούν ελευθερία της έκφρασης και ανεξιθρησκεία και άλλα σημαντικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Στοκιχόλμης. Οι δράσεις που προβλέπονται για την εφαρμογή του δείχνουν επίσης ότι πρέπει να υπάρξει συνέπεια μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνει η Ένωση και οι χώρες μέλη της με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δράση που προκύπτει από τις διεθνείς της υποχρεώσεις, παραδείγματο χάρη την ανάγκη να συμπεριληφθούν και τα θύματα βασανισμών και βασανιστήριων κατά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και ο σεβασμός της αρχής non-refoulement ή ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδών όπως αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα δράσης για τα ασυνόδευτα παιδιά. Ασυνόδευτους ανήλικους το λέει επισήμως. Υπάρχουν και άλλες πιο θεσμικές πτυχές του προβλήματος για τη μεταφορά των προβλεπομένων στην πράξη. Καταρχάς, η Κομισιόν φυσικά θα παίξει ένα ρόλο κλειδί και το έχει δείξει και προηγουμένως στην προηγούμενη περίοδο με σημαντικές προτάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα για το άσυλο ή για την ίση μεταχείριση θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μας για την εργασία της Κομισιόν στο θέμα αυτό και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει να διαπραγματεύεται για την καλύτερη εφαρμογή των προβλέψεων αυτών ακόμη και αν υπάρχουν δυσκολίες που θέτουν ορισμένες χώρες μέλη. Και είναι επίσης σημαντικό εφόσον ισχύει η χάρτα όλες οι νομοθετικές προτάσεις να αξιολογηθούν και από την άποψη των δικαιωμάτων με χαρά άκουσα από την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ ότι όντως προετοιμάζεται κάτι τέτοιο. Η αξιολόγηση αυτή βέβαια θα πρέπει όχι μόνο να σημαίνει το σεβασμό της χάρτας αλλά και των διεθνών προτύπων. Αν υπάρχει κάποια πρόταση που αφορά τα παιδιά ας πούμε πρέπει να προσέξουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδών. Δεύτερον, Ευξημένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και αυτό μια μοναδική ευκαιρία για την αύξηση της συνέπειας και της συνοχής μεταξύ των ε, προγραμμάτων της Ένωσης και των υποχρεώσεών της που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτον, θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη προοπτική στην ενδυνάμωση του ρόλου αυτής της ειδικής υπηρεσίας για για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και θα μπορέσει έτσι να επιτηρεί καλύτερα στην πράξη την εφαρμογή όχι μόνο της χάρτας αλλά και των διεθνών συμβάσεων που υποχρεώνονται να τηρήσουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό υποστηρίζουμε στεναρά την ενδυνάμωση της εντολής της και η ενδυνάμωση γενικότερα των διεθνών οργάνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που φανερά χρειάζεται να βελτιωθεί. Χρειάζεται κάποια εναρμόνιση προς τα πάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσόρ και τώρα θα ακούσουμε τον καθηγητή Στέφανο Ροντοτά. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, καιρός να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ξεπερνώντας αντιστάσεις ή εχθρότητες κάποιων πολιτικών ή την δυσπιστία και την καχυποψία κάποιων ακαδημαϊκών. Την έλλειψη ευαισθητοποίηση επίσης ορισμένου μεγάλου μέρους θα έλεγα τη κοινή γνώμη. Ο πρώτος λόγος να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας ε, τον ε, χάρτη είναι προφανής. Είναι πλέον νομικά δεσμευτικός. Δεύτερος λόγος. Αν δει ε, την ιστορική αναδρομή για το χάρτη. Και υπάρχει ένας τρίτος λόγος πολιτικός, ότι αυτός ο χάρτης είναι το επιστέγασμα μιας διαδικασίας που έχει καταστήσει την Ευρώπη, την περιοχή του κόσμου που έχει τη μεγαλύτερη προστασία για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Συνεπάγεται μια ειδική συγκεκριμένη ευθύνη για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πρώτα απ' όλα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να δουν τα θεσμικά όργανα ποιον ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο σύμφωνα και με τις τελευταίες λέξεις του προημίου του χάρτη, που λέει ότι ο χάρτης φέρει, ε, συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα σε σχέση με τους ηλικιωμένους, με την ανθρώπινη κοινωνία και τις μελλοντικέ γενιές. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ίδια νομική ιστορία του χάρτη δεν ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, θα πρέπει να θυμόμαστε τουλάχιστον ότι το Ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο κάνει δική μνήα στο χάρτη ακόμη και πριν την επίσημη διακήρυξή του στην Νίκαια το Δεκέμβριο του 2000. Το δικαστήριο τελικά αναφέρεται και αυτό στον χάρτη ως νομική βάση των αποφάσεών του. Αυτή λοιπόν η στάση είναι μια στάση στην οποία συμμερίζονται πάρα πολλές ε, αποφάσεις ε, των συνταγματικών και άλλων χαμηλόβαθμων, πιο χαμηλόβαθμων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι από το Δεκέμβριο 2000 έως το Δεκέμβριο 2009, σε αυτή τη δεκαετία, όταν συχνά σιγούσαν οι πολιτικοί, η δημιουργία της Ευρώπης ε, των ε, ελευθεριών και των δικαιωμάτων ήταν στα χέρια των δικαστικών. Τι έγινε λοιπόν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αμέσως μετά τη διακήρυξη, μετά την ανακοίνωση συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από το Βιτορίνο το Φεβρουάριο του 2001 η οποία εισάγει και ρυθμίζει την ανάγκη αξιολόγησης της συμβατότητας μεταξύ οποιοδήποτε ρυθμιστικού μέσου και του χάρτη. Αυτή η υποχρέωση πλέον έχει τηρηθεί, έχει πληρωθεί και έχει πλέον ο χάρτης καταστεί αναπίσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η συμμόρφωση λοιπόν στο χάρτη είναι προϋπόθεση για να είναι νομί, νόμιμα τα διάφορα, οι διάφορες νομοθετικές πράξεις. Αυτές, αυτή όμως η συμβατότητα με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε πολλές περιπτώσεις ήταν απλά και μόνο μια τυπική αξιολόγηση. Για να δούμε πολύ απλά ότι υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις μεταξύ του περιεχομένου ορισμένων οδηγιών και της υποτιθέμενης συμμορφωσής τους με το χάρτη. Πρέπει να συναγάγουμε από αυτό ότι ο χάρτης λαμβάνεται πιο σοβαρή υπόψη από τους δικαστές παρά από τους ε, νομοθέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως είναι καιρός ε, αυτό το χάσμα να μειωθεί. Μια ρεαλιστική προσέγγιση δείχνει ότι αν δούμε την διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και το ρόλο που θα η λεγόμενη παγκόσμια κοινότητα των δικαστηρίων. Θα δούμε ότι ο ρόλο αυτό είναι σημαντικό και θα είναι ακόμα σημαντικότερο στο μέλλον. Και αυτή την ε, εντύπωση, αυτό το συμπέρασμα το επιβεβαιώνει και η εμπειρία μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δικαστικοί μπορούν να ή να ε, εκδεθούν κάποιων εμφυδνών που έχουν. Ο χάρτης παράγει, προβλέπει και παρέχει ένα νέο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από το αδιέρετον των δικαιωμάτων. Και είναι ένα απόδραστο χαρακτηριστικό του χάρτη, που όμως η λογική της αγοράς και οι παράμετροι ασφαλείας το θέτουν υπό αφισβήτηση συνεχώς. Και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα ιεραρχία που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τους λόγους για τους οποίους ε, συντάχθηκε ο χάρτης. Μια σημαντική δήλωση στο προήμιο λέει ότι ο χάρτης τοποθετεί το πρόσωπο, το άτομο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του. Οικονομική ελευθερία δεν μπορεί να είναι μια ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία θα επιβάλλει τις ε, δικές της ανάγκες όλα τα άλλα δικαιώματα. Ακόμη και σε καιρούς κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Όταν υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες με στόχο να θυσιαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να θυμόμαστε την εντολή του Συμβουλίου της Κολονίας το 1999 που εκκίνησε, που μάλλον τη διαδικασία της ε, θεσμοθέτησης χρειάζεται για την ίδια την νομιμότητα, την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός ο χάρτης. Αυτό περιλαμβάνεται στην εντολή, δηλαδή δεν αρκούσε η νομιμοποίηση των αγορών. Χρειάζεται νομιμοποίηση μέσω δικαιωμάτων για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρη νομιμότητα και νομιμοποίηση. Ίσως θα θυμάστε τι λέει το άρθρο 19 της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη μια κοινωνία όπου δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών και όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται, δεν πρόκειται για μια συνταγματική κατάσταση. Θα πρέπει να υπερβούμε ε, την, ε, θεώρηση, την υπερβολική θεώρηση της αγοράς. Δεν θα πρέπει να γυρίσουμε προς τα πίσω. Πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία που θα αντικατοπτρίζει την ασυνέχεια η οποία έχει εισαχθεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα από τη σύγκληση ελευθεριών δικαιωμάτων προσώπων. Το ερώτημα είναι το εξής. Η ελευθερία υπό την πλήρη της έννοια μπορεί να επιβιώσει σε μια εποχή όπου οικονομικές δυσκολίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα ή ως πρόφαση, ως πρόσχημα για τον περιορισμό των ελευθεριών αυτών. Ερχόμενος ε, στα ζητήματα της ασφάλειας, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις. Στις 2 Μαρτίου του τρέχοντος, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε ότι είναι ασυμβίβαστο με τη συνταγματική νομική ταυτότητα της, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας η Ευρωπαϊκή Οδηγία 24 το 2006. Λέει λοιπόν το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Bundesverfassung Gerecht, ότι η προστασία δεν περιλαμβάνει μόνο το περιεχόμενο και άλλα στοιχεία ε, που έχουν να κάνουν με το απόρριτο. Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ε, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα για διάφορα στρώματα της ιδιωτικής σφαίρας, της ιδιωτικής ζωής ε, του ανθρώπου. και κάποια άλλα πράγματα λοιπόν που λέγονται στην απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου που κατελικά καθιστούν να συμβίβαστη την ε, οδηγία της συγκεκριμένη. Παράβαση της ελευθερίας ε, των ανθρώπων αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του χάρτη για την ε, Συμφωνία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς λοιπόν θα αντιδράσουν στην απόφαση αυτή οι Ευρωπαίοι νομοθέτες. Είχαμε κάποια πρόσφατα δείγματα που δυστυχώς δεν ε, προσφέρονται για ιδιαίτερα αισιοδοξία. Υπάρχει ένα έγγραφο του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου για τα μέσα συγκέντρωσης δεδομένων και πληροφοριών για διαδικασίες βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Και εκεί αναφέρονται 70 ερωτήματα για να διαγραφεί, να σκιαγραφηθεί το προφίλ κάποιων προσώπων, στιγματοποίηση περιφορών, κατάταξη, ταξινόμηση ανθρώπων λόγω ιδεολογίας προσωπικών σχέσεων κτλ. κτλ. Διατρέχουμε τον κίνδυνο οι κοινωνίες μας να γίνουν έθνη υπόπτων όπου θα παραβιάζεται τελικά ο χάρτης, θα παραβιάζονται ελευθερίες, ελευθερίας έκφρασης και τα λοιπά. Και συνεταιρίζεστε. Έτσι κινδυνεύουμε να νομιμοποιήσουμε το ψηφιακό τσουνάμι που μπορεί να επακολουθήσει ως αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών. Και ιδίως μέσω του διαδικτύου. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο να αντιδράσει ή μήπω πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει παρέμβαση από κάποια δικαστήρια που θα επιβεβαιώνουν ότι προστασία δικαιωμάτων και ελευθερών στην Ευρώπη μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από το δικαστικό σώμα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ο χάρτης είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ατού. Πολλοί και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο που μπορεί να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να έχει μια παγκόσμια επιρροή το βλέπουν ιδιαίτερα θετικό μάτι. Η δύναμη της ελευθερίας είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσουμε. Σας ευχαριστώ. Professore. Ολοκληρώσατε καθηγητά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ποιος είναι ο θέλει να λάβει το λόγο? Η κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ομιλίες που έγιναν Έχω ωστόσο κάποιες παρατηρήσεις να κάνω σε αυτά που ελέγχθησαν. Όταν ε, δουλεύαμε για την ε, εντολή προς την, ε, για την υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βιέννης είχαμε εκφράσει κάποιες επιθυμίες ως κοινοβούλιο και είχαμε μιλήσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα και πραγματικά θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό σημαντικό η υπηρεσία αυτή να δίνει και να μας δίνει και σωστά στοιχεία και δεδομένα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τους τρόπους και τα μέσα να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αυτά γιατί πιστεύω ότι και το Κοινοβούλιο και άλλοι φορείς θεωρούν ότι η υπηρεσία της Βιέννης κάνει πολύ καλές εξέσεις όμως οι εξέσεις αυτές δεν μπορούν άμεσα να συνδυαστούν με τη δουλειά μας. Η υπηρεσία λοιπόν φαίνεται να δουλεύει σαν ερευνητικό κέντρο κατά κύριο λόγο και όχι έτσι όπως θυμούσαμε εμείς. Όταν λοιπόν προχωρήσουμε σε ένα θεώρηση της εντολής για την υπηρεσία της Βιέννης θα πρέπει να τα σκεφτούμε ξανά αυτά τα πράγματα και να είμαστε σαφέστεροι. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της υπηρεσίας αυτής εφόσον η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δεσμευτική ήταν σαφή ο ρόλο τη υπηρεσία πριν όταν η χάρτα δεν ήταν νομικά δεσμευτική τώρα βεβαίω ενισχύεται ίσως ο ρόλος της υπηρεσίας θεωρώ ότι σημαντικό θα ήταν η υπηρεσία αυτή να ασχοληθεί με τα θέματα που έθεσε ο κύριος Τζάραμπ θα μπορούσε η υπηρεσία να είναι ο φορέας, ο οργανισμός που θα συνδέει τα διεθνή πρότυπα τα οποία ακολουθούν και κάποια κράτη-μέλη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αν θέλετε και μπορούσε και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα στην παρακολούθηση αν θέλετε για τη συμμόρφωση από πλευρά κρατών μελών. Είναι, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η υπηρεσία αυτή ο οργανισμός να συνεργαστεί στενά και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία και των μεν και των δε σωστά. Διότι πρέπει να υπάρχει να συνδυαστούν και να συγκριθούν αν θέλετε τα πρότυπα τα, της Ευρώπης με αυτά του υπόλοιπου κόσμου και των διεθνών οργανισμών. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπε ο κύριο πράγματι πρέπει να παρακολουθούμε, να αποπτεύουμε την εφαρμογή, να δούμε πώς αν υπάρχει συμμόρφωση ή όχι και βεβαίως θα θυμάστε ότι στην τελευταία συζήτηση που κάναμε για ανθρώπινα δικαιώματα στην Ολομέλεια είχα ρωτήσει εγώ την κυρία Άστον για το πώς θα καλυφθεί και ο τομέας αυτός από την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερική δράση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, ο Ντέιβιτ Σκίνερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ, ναι, πρόεδρε. Εδώ εκπροσωπούμε δέκα εθνικές μήκη όμικρον. Έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, το νόημα και τη σημασία της ενίας της αντιρρήσης συνειδήσεως που το αναφέρει το άρθρο 10 για την ελευθερία συνείδησης και την ανεξιθρησκεία. Στα αγγλικά λέει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης αναγνωρίζεται σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους που την διέπουν. Γενικά όμως εννοούμε ότι πρόκειται για αντίρρηση της στρατιωτικής θητείας ενώ στα γερμανικά γίνεται και συγκεκριμένη μνήμα ότι το δικαίωμα αυτό χρησιμοποιήθηκε στους παγκοσμίους πολέμους. Στα αγγλικά όμως δεν το λέει, είναι πιο γενικό. Εφόσον ζούμε σε εποχή όπου συνυπάρχουν πολλές μειονότητες, αυτό το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης που αναφέρει ρητά η χάρτα θα μπορούσε να εφαρμόζεται και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στη στρατιωτική θητεία. Μπορεί κάποιος να θέλει να ασκήσει οποιοδήποτε τμήμα της συνείδησης του. Ας πούμε μπορεί μερικοί να αρνούνται την μερικοί γιατροί να αρνούνται να κάνουν εκτρώσεις. Οι γονείς μπορεί να ζητήσουν εξαίρεση από θρησκευτική στρατιωτική εκπαίδευση και άρα αυτό ανοίγει την πόρτα σε πολλά. Εμείς θεωρούμε ότι αν κάποιος ή κάποιοι έχουν ορισμένες ισχυρές πεπιθήσεις που είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν για αυτές, τότε το δικαίωμα αυτό στην ε, αντίρρηση συνείδησης είναι σωστό να θεωρείται σεβαστό, αλλά ερωτούμε, ερωτούμε ιδίω ιδιαίτερα τον κύριο Ρεντόλτο που συνεισέφερε στη συγγραφή της χάρτας, ερωτούμε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το τμήμα 2 του άρθρου αυτού, το εδάφιο 2, εάν χρειαστεί θα μπορούσε να επεκταθεί και σε θέματα πέραν της στρατιωτικής θητείας και σε τομείς που αφορούν γενικότερα θρησκευτικά, φιλοσοφικά, ανθρωπιστικά θέματα. Γιατί πολλές μήκοι όμικρον ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Όσο συζητιέται περισσότερο ως δεσμευτικό εργαλείο η χάρτα. Και εδώ πρόκειται ίσως για θεμελιώδεις όντως ελευθερίες που πρέπει όμως να αποσαφινιστούν. Δεύτερο ερώτημα στον διευθυντή Φρά. Πριν από μερικά χρόνια ήρθαμε σε μία ακρόαση εδώ στις Βρυξέλλες και θυμάμαι ότι είχε πει τότε ότι δεν είναι σε θέση να παρέμβει ή να αναλάβει περιπτώσεις απλώς επιτηρεί και γράφει μια ετήσια έκθεση Τώρα που αυξάνονται οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπά Δεν θα μπορούσε η υπηρεσία αυτή να επεκταθεί και αυτή ώστε να ελέγχει και άλλες περιπτώσεις παραβίασης της χάρτας και να έχει περισσότερη δικαιοδοσία να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σκίνερ. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ερώτημα αυτό που θέλω να θέσω, αλλά είναι μία δήλωση που τη θεωρούμε σημαντική για τη συζήτηση. Εκτός από όσα υπόθηκαν σήμερα από την κυρία Ρέντινγκ και για, τις υπο, για, για όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, η Κομισιόν χρηματοδοτεί και ανεξάρτητες έρευνες και μελέτες, σύμφωνα με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το τρέχον δηλαδή, και για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικο-οικονομικές αναφέρονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όχι μόνο ο χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα στο σύνολο του κόσμου. Διασφαλίζουμε οι μελέτες και έρευνες αυτές φυσικά να συμφωνούν και εσωτερικά με τις νομοθετικές διαδικασίες και με τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς συμβάσεις. Αλλά θεωρούμε ότι η έρευνα αυτή θα ενδιέφερε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου να γνωρίζουν δηλαδή τα αποτελέσματα των μελετών και ερευνών αυτών. Αν χρειαστούν περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ να ρωτήσετε την Επιτροπή και δεν θα διστάσει να σας απαντήσει. Νομίζω ότι έπρεπε να σας τα πω αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, λέει ο πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν να θέλει το λόγο, οπότε επανέρχομαι στους ομιλητές Τζάραμπ, Ροντουτά, ετέθησαν ερωτήσεις προς εσάς προσωπικώς, οπότε ακούμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις και τα σχόλια που έγιναν. Άκουσα ένα πολύ σημαντικό ερώτημα σχετικά με το ο, πότε και πώς κάνουμε τις μελέτες μας και πώς αυτά συνδέονται με τη δική σας τη δουλειά. Είναι πραγματικά ένα καλό παράδειγμα είναι το πρόσφατο, η πρόσφατη έρευνα για την ομοφοβία, ομοφιλοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, ε ακριβώς τη στιγμή που υποβάλλονταν η έγκριση του σχέδιου οδηγίας υποβάλλαμε και εμείς την εκθεσή μας. Τέτοιου είδους συντονισμός ε, δράσεων θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να γίνει καλύτερα στο μέλλον. Πράγματι έχουμε στενή επαφή με την Επιτροπή σας και ε, όντως θα θέλαμε να δούμε ακριβώ ποιο είναι το δικό σας χρονοπρόγραμμα για να το συνδυάσουμε με το δικό μα. Βεβαίω, πέρα από την ομοφιλοφοβία ε, ασχοληθήκαμε και άλλα, ε, με άλλα θέματα όπως παραδείγματος χάρη τα συνόδευτα παιδιά ε, που ζητούν άσυλο αυτά τα κάναμε σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν εδώ αλλά αυτά όλα πρέπει να ενισχυθούν μας ενδιαφέρει να φτιάχνουμε καλές εξαίσεις με βάση αντικειμενικά στοιχεία. Αλλά βεβαίως αυτό είναι ο ένας στόχος μας. Ο άλλος στόχος μας είναι να συνδυαζόμαστε και με ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και τα λοιπά ώστε να επηρεάσουμε, να επηρεάζουμε και την πολιτική που χαράζεται στην Ένωση. από τις ε, συναντήσεις που κάναμε με, με ε, τώρα έχουμε πολλά ε, ακόμη να σκεφτούμε και Βεβαίω υπάρχει πέρα από το συντονισμό και συγχρονισμό των προσπαθειών μας και το θέμα του της δημοσιοποίησης αν θέλετε των εξαίσεων αυτών πιο ε, επικοινωνιακά τι πρέπει να κάνουμε για να είναι και προσβάσιμες οι εκθέσεις μας από τον Ευρωπαίο πολίτη και από όλους Καταλαβαίνω βέβαια και την παρατήρηση που έγινε που έκανε και ο Τζαν, Γιάν Τζάραμπ το συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πράγματι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, λαμβάνονται υπόψη και συνδυάζονται με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης. Όταν φτιάξαμε την έκθεση για τα συνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο, χρησιμοποιήσαμε σαφέστατα συμβάσει των Ηνωμένων Εθνών, τα δικαιώματα των παιδιών των Ηνωμένων Εθνών, σχετική χάρτα και κάποιες εθνικές συμβάσεις πλαίσιο για τις εθνωτικές μειονότητες. Υπάρχουν πολλά λοιπόν ε, που μπορούμε ακόμη να κάνουμε. Και βεβαίω θυμίζω εδώ και την κατευθύνια γραμμή 5 που ανέκριναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και που ουσιαστικά εισάγουν αν θέλετε στο ενωσιακό πλαίσιο τα στάνταρτ, τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα για τους αντιρρησίες συνείδησης. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά θα το αφήσω, θα αφήσω να το ε, επεξεργαστεί ο κύριος Ροντοτά. Τώρα, να πω εγώ τώρα ότι υπάρχει και ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που φτιάχτηκε πριν από 4-5 χρόνια και το δίκτυο αυτό εκπώνησε μια γνωμοδότηση, αν μπορώ να την πω έτσι, για τα αυτά που είπατε και ιδιαίτερα για τον ιατρικό τομέα. Σε ποιο βαθμό δηλαδή ο γιατρός θα μπορούσε να επικαλεστεί την συνείδησή του για να αρνηθεί να κάνει μια απόξεση και όχι μόνο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια διάταξη που λέει ότι ότι στον οργανισμό μας που λέει ότι ε, εάν συμβαίνει, αν συμβεί ένα πολύ σοβαρό γεγονός μπορούμε να εκπονήσουμε έξεση για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός αυτό έγινε στο παρελθόν αλλά οι κανονισμοί είναι αρκετά περιορισμένοι όσον αφορά το δικαίωμα πρωτοβουλίας μας αν θέλετε Άρα έχουμε και περιορισμένες αρμοδιότητες για την εποπτεία και τον έλεγχο. Ε, ωστόσο, θέματα σαν και αυτά πραγματικά της αντίρρησης συνείδησης είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει να συζητηθούν και στον οργανισμό μας υπάρχει και το ενδεχόμενο αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού ε, οπότε μπορεί τότε να ε, σκεφτούμε αν πρέπει να περιλάβουμε σε αρμοδιότητες κάποια τέτοια πράγματα. Αυτό θα γίνει λόγω μετά από την πενταετία ζωής που έχει ο οργανισμός μας πια. Τζάραμπ. Ας κάνουμε θα ήθελα να μπορούσα να κάνω πιο ζωντανή τη συζήτηση ε, δηλώνοντας αντιρρήσεις για κάποια πράγματα που ελέγχθησαν αλλά δυστυχώ δεν μπορώ συμφωνώ με όλα αυτά που ελέγχθησαν η συνέπεια ε, των δικών μας προτύπων με αυτά άλλων διεθνών οργανισμών Συμβουλίου της Ευρώπης κτλ. είναι απαραίτητη. Και βεβαίως αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν δουλεύουμε με τη χάρτα που είναι βέβαια το κύριο εργαλείο μας. Ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βιέννης είναι ο πιο ενδεδειγμένος για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά αλλά και με άλλους φορείς, με το κοινοβούλιο, με τους, τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκινάει τις ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροντώτα Μερικά σύντομα, σύντομα για την αντίρρηση συνειδήσεως. Το δικαίωμα αυτό έχει αναφερθεί με τρόπο γενικότερο όχι μόνο θρησκευτικό και για τη στρατιωτική θητεία. Είναι φανερό ότι ξεπερνάει την παραδοσιακή έννοια που είχε δοθεί για αντίρρηση στη στρατιωτική θητεία. Το ουσιώδες εδώ είναι στις τελευταίες λέξεις του τμήμα του εδαφίου 2 του άρθρου αυτού. Λέει σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Και γιατί το βάλαμε αυτό αυτή τη διατύπωση. Γενικά διότι υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες ανάλογα με τη χώρα. Σήμερα το ενδιαφέρον είναι το ουσιώδες ότι η παραδοσιακή η συνήθις αντίρρηση στη στρατιωτική θητεία δεν είχε επίπτωση επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των λαών. Δηλαδή, αν είστε γιατρός και έχετε αντίρρηση στις εκτρώσεις ή στη χορήγηση χαπιών που εμποδίζουν τη σύλληψη, αντισυλληπτικών δηλαδή. Έχετε επιπτώσεις τότε στο δικαίωμα της γυναίκας να έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες και μπορεί αυτό να οδηγήσει σε δύο λύσεις. Πρώτον, αποκλισμός, άρνηση δηλαδή του δικαιώματος αντίρρησης ή για την αντίρρηση στις εκτρώσεις, ο Ιταλικός νόμος λέει ότι διό, επειδή η έκτρωση είναι νόμιμη μόνο μέσα στις δημόσιες δομές, έχει δικαίωμα ο γιατρός να εκφράσει αντίρρηση και υποχρέωση το νοσοκομείο ούτως ή άλλως να χορηγήσει την υπηρεσία στις γυναίκες που τη ζητούν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι στην πρόθεση του νομοθέτη πρόκειται για γενικότερο δικαίωμα που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς. Αλλά επειδή το πρόβλημα αυτό προερχόταν από από την αντίρρηση eh, στον πόλεμο χρειάστηκε η διευκρίνηση. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί η αντίρρηση συνειδήσεως για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως τους δικαστάς να γίνει αποδεκτή. Να γίνει αποδεκτή. Α, ο κύριος Σκίνερ νομίζω θέλει να απαντήσει. Ορίστε παρακαλώ. Αλλά σύντομα, σύντομα, σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα, συντομότατα. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος πως ότι έχει ευρύτερη σημασία το δικαίωμα αυτό, γιατί τότε στη γερμανική μετάφραση περιορίζεται στη στρατιωτική θητεία. Υπάρχει εδώ μια ασάφεια. Ορίστε. Θέλει κανείς να απαντήσει, μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Μήπως ο κύριος Γκέροπ. Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω τη γερμανική μετάφραση. Αλλά στις υποσημειώσεις της χάρτας βλέπετε ότι υπάρχει μια εξήγηση που σας είπα προηγουμένως. προηγουμένως. Α, τότε καλά. Κανένα άλλο σχόλιο, καμία άλλη ερώτηση, όχι, τότε καλά. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η συζήτηση για τον χώρο ασφαλείας. Έχουμε κι άλλους εδώ μιλητάς που μας κάνουν την τιμή να έχουν προσέλθει και πρώτος και καλύτερος ο κύριος Ανρί Λαμπίλ, Λαμπέλ που είναι καθηγητής της νομικής σχολής της Μπαγιών Πανεπιστήμιο Πάου και των περιοχών Αντούρ γύρω από το ποτάμι Αντούρ και μετά θα ομιλήσει ο κύριος Μιχαήλ Πριβό, διευθυντής του ΕΝΑΡ και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της τρίτης πλατφόρμας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και στο, μετά ο κύριος Έμον Άοντα, Γενικό Διευθυντή τη Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ομάδα Εθνικών Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο κύριο Δαβίδ Νίκολς ασκών καθήκοντα διευθυντή του Γραφείου Διεθνούς Αμνηστίας της ΕΕ. Προτείνω να ακούσουμε τους ομιλητάς για 8-10 λεπτά τον καθένα και μετά να αρχίσουμε την τελευταία μας συζήτηση πριν λήξει το σεμινάριο. Πρώτος είπα και καλύτερος ο κύριος Ανρί Λαμπέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι βέβαια ιδιαιτέρως που μπορώ εδώ να μιλήσω για την επίπτωση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και για μια σειρά από λόγους, πρώτος εκ των οποίων βέβαια είναι ότι προκαλεί κάποιο είδους έκπληξη και απορία να βλέπει κανείς σήμερα κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της συνθήκης της ε, Λισαβόνας να περνά σε ίσως σε δεύτερο πλάνο τη ανησυχία και του ενδιαφέροντος όταν μιλάμε για την ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Καταρχάς πρέπει να επενθυμίσουμε ότι Έχουμε ήδη περάσει ε, ε, μια δεκαετία ε, με σημαντική πρόοδο και ίσως ανέλπιστη θα μπορούσε να πει κανείς για αυτό το χώρο. Πρώτος, πρώτη δεκαετία λοιπόν του χώρου ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας χωρίς να έχουμε όμως κάποια πράξεις αναφοράς, θεμελιώδες δίκαιο δηλαδή, χωρίς κάποια ρυθμιστικά, κανονιστικά ερίσματα. Οπότε τότε οι δικαστές δεν είχαν κάποια σημεία αναφοράς, δεν είχαν ένα εργαλείο όπως αυτό που είναι η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να αναφέρονται. Θεωρώ λοιπόν λίγο περίεργο τον, μη, τον ελάσσονα ρόλο που φαίνεται να έχει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τότε που ουτέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, θα θυμάστε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις ε, για την ε, συνθήκη η υπήρξαν κάποια σημεία διένεξη, μεταξύ αυτών ήταν ο χάρτη μιλητών δικαιωμάτων. Και κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματικά είχαν προσπαθήσει επανειλημμένω να αποσταθεροποιήσουν αυτό το οποίο είχε εγκριθεί στην Νίκαια το 2000, επί Γαλλικής Προεδρίας τότε. Και το τελικό αποτέλεσμα της συνθήκης της Λισαβόνας ήταν τελικά ότι κρύφτηκε, αν θέλετε, συγκαλύφθηκε σε ένα παράρτημα και όχι σε ένα δεύτερο τμήμα συνταγματική συνθήκη Αυτό, ο χάρη των δικαιωμάτων. Φάνηκε λοιπόν να δίνεται προτεραιότητα σε αυτό που θεωρήθηκε ως η μεγάλη καινοτομία, δηλαδή η προοπτική ένταξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προβολείς έχουν κυρίως επικεντρωθεί σε αυτό, στην προσχώρηση της Ένωσης, στην ε, διαπραγματευτική εντολή και όχι τόσο στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποτελέσει η χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Απορρέει λοιπόν από όλα αυτά Μία κάπως μινιμαλιστική ε, παρουσίαση του χάρτη μελίων δικαιωμάτων στην κοινή γνώμη που κατά κάποιο τρόπο θεωρείται λίγο ε, κάτι τετριμένο. Ότι δηλαδή δεν φέρνει και κάτι το τόσο πολύ καινοτόμο και σημαντικό ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για τα κράτη-μέλη σαν απλά να περιοριζόταν στην ε, συνταγματοποίηση ή στην εγγραφή ε, στο συνθήκη, στο κείμενο, πράγματα τα οποία ήδη υπήρχαν και τα οποία ήδη ήταν αντικείμενο προστασίας. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό σφάλμα. Είναι ένα σοβαρό σφάλμα πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την αξία του χάρτη. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ποια είναι η αξία του πρωτογενούς δικαίου, δηλαδή των συνθήκων. Είναι σημαντικό το λάθο λοιπόν και ω προ το περιεχόμενο, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναπτύσσει μια σειρά δικαιωμάτων τα οποία σήμερα δεν περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν είναι και γνωστά σε κάποια κράτη-μέλη. Μιλήσαμε πριν για την προστασία δεδομένων, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα δικαιώματα ηθαγένεια, το δικαίωμα για την καλή διαχείριση δίκη κτλ. Για πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα υποχρεώσουν την Ένωση και τα κράτη-μέλη να εργαστούν διαφορετικά. Άρα, νομίζω ότι σήμερα ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει πραγματικά να ε, αντιμετωπιστεί ως αυτό που είναι πραγματικά. Γιατί το πρώτο λάθος είναι να θεωρεί κανείς ότι το κείμενο αυτό δεν αποτελεί κάτι καινούριο. Το κείμενο αυτό, επενθυμίζουμε, είναι δεσμευτικό από νομικής πλευράς και μπορεί κανείς να ε, κάνει αναφορά και επίκλησή του και στα εθνικά και στα κοινοτικά δικαστήρια. Και αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον ε, εξ όσων εγώ κρίνω. Ο χάρτης είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι διατρέχει και διαπνέει όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε βρίσκεται και στο μάτι του κυκλώνα, γιατί δεν υπάρχει άλλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να ενδιαφέρεται τόσο πολύ ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι σαφέ ότι ο χώρο ασφάλεια, δικαιοσύνη και ασφάλεια είναι ακριβώ ο πρώτος ε, που θα φυγεί, αν θέλετε, από, και που αφοράται από αυτό ε, την δεσμευτική ισχύ του χάρτη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί κανείς να εμείνει ε, να κάνει αυτά που έκανε στο παρελθόν. Δεν είναι ένα απλά θυμοτυπικό ε, που μπαίνει δηλαδή το άρθρο, σε οποιοδήποτε άρθρο ή αναφορά στο χάρτη όπως π.χ. Ε, είναι η ρήτρα για την επικουρικότητα. Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει σήμερα να δεχθούμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα συνεπάγονται μια εγκάρσια ματιά η οποία δηλαδή διατρέχει όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται σε, στο σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Άρα, για μένα αυτό συνεπάγεται σημαντικούς περιορισμούς. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καινούργοι για τα διάφορα θεσμικά όργανα και για τα λίγα λεπτά που μου απομένουν θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο σημεία θα αναφέρω είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δικά της, ε, το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί. Δεν δείχνει τελικά να θέλει να βάλει στο επίκεντρο των δράσεών του τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως ό,τι αφορά αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή όμω οι δύο τομεί, ο νομοθέτης και ο δικαστή ε, της Ευρωπαϊκής για αυτού θέλω να μιλήσω κυρίω. Νομοθέτη πρώτα και πώ επηρεάζει ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τον νομοθέτη παρά την εξαιρετική μετάβαση που είχαμε σε ό,τι αφορά το χώρο ελευθερία ασφάλεια δικαιοσύνη με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, παρά λοιπόν τη μετάβαση στην κοινοτική μέθοδο και στη συναπόφαση και στον κανονικό έλεγχο, τακτικό έλεγχο του δικαστή, κοινά δικαιώματα κτλ. Έχουμε παρόλα αυτά το, την εντύπωση ότι δεν όχι απλά δεν έχουν, δεν αλλάξει τα πράγματα, όλα ότι παραμένουν και ω είχαν. Δηλαδή, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ναι μεν ε, θεωρείται κάτι θετικό, αλλά αντιμετωπίζεται με παθητικό τρόπο. Και τελικά έχουμε ένα κατάλογο, ε, αυτός είναι δηλαδή ο χάρτης, ένας κατάλογος ε, που με τα ευλαβία ευλαβία ε, τον ξεφυλίζουμε και τον αναφέρουμε όποτε μπορούμε όπως παλιά είχαμε κάποιες, ε, ε, κάποιες υποχρεωτικές φιγούρες ε, στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Αλλά υπήρχαν και κάποιες άλλες ελεύθερες φιγούρες. Εδώ έχουμε την εντύπωση ότι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι σαν ένα μήνυμα που στέλνουμε ότι ορίστε η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και μετά όταν έρχεται η στιγμή να ανοίξουμε το φάκελο με τα πραγματικά θέματα, αυτόν τον βάζουμε κατά μέρο. Υπάρχει εδώ κατά την άποψή μου ένας κίνδυνος ο οποίος απειλεί, πώς να σας το πω, την ε, άνθηση, την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χάρτη. έχω φτάσει εδώ ε, διασχίζοντας τη Γαλλία. Δεν ε, μιλώ με υπονοούμενο ούτε με υπεκφυγές, θα έχετε καταλάβει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσουμε για την τεχνοκρατική προσέγγιση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Εδώ και πολύ καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λέμε και επαναλαμβάνουμε τη φράση impact assessment, αξιολόγηση επιπτώσεων. Μα δεν έχει γίνει. Ε, Παραδείγματο χάρη για την οδηγία για την οικογενειακή επανένωση. Όταν ε, θέλαμε να, περάσουμε, να περάσουν από κάποιε εξετάσει τα παιδιά για να βρουν ε, του γονεί του, για να επανενωθούν την οικογένειά του. Δεν υπήρχαν κάποιε ε, διαφορέ και διαμάχε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα μπορούσε να πει κανεί ναι, τα λύσαμε, τα διευθετήσαμε και προχωράμε. Όχι όμω. Δεν έχει γίνει αυτό. Πρώτη λοιπόν, πρώτος κίνδυνος, τεχνοκρατική προσέγγιση. Δεύτερος κίνδυνος, μία αγγελική, αν θέλετε, προσέγγιση. Μπορεί τελικά να φτάσουμε χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις εκφράσεις c'est le plus sûr moyen de ne pas permettre de les respecter στην έννοια του ανθρωποδικαιωματισμού. Υπάρχει μια άρνηση λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή ε, του να δούμε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι με αυτά τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Βλέπω ότι υπάρχουν δύο προκλήσεις, ε, δύο ειδών προκλήσεις, τεχνικές και πολιτικές. Μια τεχνική πρόκληση. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφέρει από την έλλειψη προληπτικών μηχανισμών. Μιλώ ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους ελλείψεις σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω προληπτικού έλεγχου της συνταγματικότητας. στην παραγωγή προτύπων πρέπει να συμπεριληφθεί ε, ο χάρτης και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνεται και ανάντι και κατάντι ο έλεγχος και θα πρέπει να προβλεφθούν μηχανισμοί για να μπορεί να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση των κειμένων που εγκρίνουμε με τις διατάξεις του χάρτη. Κάτι άλλο και σημαντικότερο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ασφάλεια Δικαιοσύνη Ελευθερία. Και επενθυμίζω ότι η ιδιαιτερότητα αυτού του χώρου είναι ότι έχουμε εδώ το δικαίωμα έμεσης εφαρμογής, δηλαδή έμεσης εκτελεστότητας. Οι κανόνες δηλαδή οι οποίοι εκπονούνται σε αυτό το χώρο είναι πράξεις που θα πρέπει συνέχεια να μεταφορθούν στο εθνικό δίκαιο ως οδηγίες. Άρα κατά τη φάση αυτή της μετάβασης κάποιες φορές υπάρχει ίσως ένα περιθώριο παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητα, την ακριβή και απόλυτη εγκυρότητα των κειμένων που εγκρίνουμε. Επίσης, ε, ως τεχνική πρόκληση, υπάρχει μια απειλή για το ουσιαστικό δίκαιο ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος βασίζεται σε μια αρχή που αναφέρεται στη συνθήκη και μια που δεν αναφέρεται. Πρώτα απ' όλα αμοιβαία αναγνώριση. Πώ να λειτουργήσει αυτή, αν δεν συμφωνούμε για το επίπεδο προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεύτερη αρχή, που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή και σε ό,τι αφορά ιδίω ε, την ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων, είναι η αρχή τη διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα εδώ όμω μπορεί να ισχύει μόνο αν τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν τον κοινό παρονομαστή που επιτρέπει την ανταλλαγή των πληροφοριών. Τρίτη τεχνική πρόκληση για τον νομοθέτη. Κάτι πολύ σημαντικό και για τους ε, φορείς ε, του χώρου αυτού ή το, το Eurojust, Just, ε, η Frontex, η Europol, όλοι αυτοί οι φορείς που εντάσσονται σε αυτό το χώρο. Πρέπει να σέβονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στο χάρτη και να τον εντάξουν. Ή υπάρχουν κάποιες άλλες εξοδοφικές δράσεις. μία περίπολος, ένα πλοίο που έχει κάποιους πρόσφυγες από τη Σενεγάλη, από τη Λιβύη τι κάνουμε με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, θα μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες υποχρεώσεις που σχετίζονται με, την, ε, με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και έτσι έρχομαι στο εξή. Από τεχνική πλευράς εδώ και επανέρχομαι ε, και θα, δω και θα σας μιλήσω για την εικόνα του δικαστή. μία από τις μεγάλες προκλήσεις για τον Λομοθέτη και για το Κοινοβούλιο θα είναι μάλλον να συλλάβει και να οικοδομήσει, να σκιαγραφίσει ε, και να φτιάξει τελικά ένα πραγματικό ιστό αράχνης, όπου σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια και με τα θεσμικά όργανα που είναι φορτισμένα ε, με την εφαρμογή κάποιων δικαιωμάτων και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Παραδείγματο χάρη, κάποιοι φορεί για την προστασία των ε, δεδομένων. Ακούσαμε τον Ευρωπαϊκό Ελεγκτή χθε. Αυτό ο ιστό τη αράχνη λοιπόν θα πρέπει να γίνει ώστε αυτά τα οποία είναι απλά και μόνο διακηρυγμένα δικαιώματα και μένουν στις λέξεις, μένουν στα λόγια, να μεταφερθούν και στις, σε πράξεις, να γίνουν έργο. Και έρχομαι στη δεύτερη πρόκληση που αφορά τον νομοθέτη. Είναι μια πρόκληση πολιτική υφή, πολιτικού χαρακτήρα. Και νομίζω ότι πρέπει, δεν πρέπει να φοβόμαστε να αναλάβουμε αυτή την πρόκληση. Πρώτα απ' όλα, πρόκληση ό,τι αφορά την αυτονομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δεχθούμε και να πούμε ξεκάθαρα, ρητά, ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένα ιδιαίτερο ε, μέσο εγκάρσιο που περιλαμβάνει νέα δικαιώματα και το οποίο θα πρέπει να μπορέσει να ανοίξει τα φτερά του αν θέλετε και να ζήσει πλήρως τη ζωή του και όχι να κρύβεται ε, πίσω από άλλα κείμενα διεθνή ε, για την προστασία δικαιωμάτων. Η κοινοτική λογική και η κοινοτική μέθοδο, μα έδωσαν τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε για 50 χρόνια μια Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση κανόνε συμπεριφορά, με βάση κοινέ αξίε. και δεν θα πρέπει να ε, διαχυθεί ε, με αυτό με βάση αυτά που έγιναν σε άλλα φόρα ε, για άλλους, για να πληρώσουν άλλους σκοπούς. Θα πρέπει λοιπόν η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιδιαίτερη θέση που έχει στον πλανήτη, να εδρωθεί και να παγιωθεί σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το είπε και ένας από τους προλαλήσαντες. Και έρχομαι στη δεύτερη πρόκληση, την πολιτική πρόκληση που είναι η διάρθρωση και η σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο προσχώρηση σε άλλα διεθνεί φορεί προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμβαση της Γενέβης μου έρχεται στο μυαλό, παραδείγματος χάρη. Μπορούμε να συνεχίσουμε επιμακρό να λέμε ότι ε, τα μέτρα που σχετίζονται με το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνάδουν, είναι σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενέβης. Η έγκριση μια παράγωγη νομοθεσία ενδεχομένω που θα εφαρμόζει τη Σύμβαση τη Γενέβη ή να μην προσχωρήσουμε σε αυτό το κείμενο που θα δημιουργήσει τεχνικά προβλήματα. Μήπω θα πρέπει να περιμένει η Κομισιόν το 2012 για να κάνει μελέτη σκοπιμότητα γιατί είναι τόσο πολύ ε, φορτωμένο το πρόγραμμά τη, αν και έχει ζητηθεί με το πρόγραμμα εργασία να γίνει ήδη από τώρα αυτή η μελέτη τη σκοπιμότητα. Ένα άλλο παράδειγμα για αυτή τη διάρθρωση και τη διασύνδεση με τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Φυσικά, είναι προφανέ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξέλθουμε από αυτή τη λογική την ιδέα ότι ο χάρτη των δικαιωμάτων τελικά είναι ένα κλόνος ένα οσία ε, τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, είναι λάθο. Πρώτον, δεν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ των δύο κειμένων. Δεν υπάρχει απόλυτη σύμπτωση μεταξύ του. Σα λέω, υπάρχουν 12 νέα δικαιώματα τα οποία δεν τα έχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λάθος επίσης γιατί η λογική των δύο κόσμων είναι διαφορετική. Είναι ένα πραγματικό θαύμα από νομολογιακή πλευρά ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έφτασε σε αυτό εξαιρετικό επίπεδο προστασία που μας εξασφαλίζει. Μπορούμε όμως πραγματικά και σοβαρά να πιστέψουμε ότι οι συντάκτες τη Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεκαετία του 50 όταν διαπραγματεύονταν το άρθρο 8 αυτή τη σύμβαση, είχαν κατά νου τα προβλήματα των δικαιωμάτων των ε, τρανσέξουαλ, των ομοφιλόφιλων, ε, των ε, παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου ή της προστασίας των δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση. Και το να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα οφείλει όλα στον δικαστή και στην ευφυΐα του δικαστή που καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα ζωντανό κείμενο και ότι θα πρέπει αυτό να ερμηνεύεται με βάση τις εξελίξεις και την πρόοδο. Και η λογική του κοινωτικού δικαίου δεν έχει καμία σχέση. Ούτε η λογική τη Ευρωπαϊκή Ένωση καμία σχέση με όλα αυτά. Ιδίω γιατί η λογική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ε, απόλυτα αληθέ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου, είναι να παράγει κανόνε, να παράγει δίκαιο, δεσμευτικό δίκαιο για του παραλήπτε του, για του αποδέκτε του. Εδώ η συλλογιστική και ο τρόπο εργασία είναι εντελώ αντίστροφο. Επομένω, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χάρτη των δημιουργικών δικαιωμάτων σχετίζεται άρρηκτα με την παραγωγή δικαίου εδώ, ε, στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίζουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκού νόμου, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη μα την ε, νομοθετική πράξη αναφορά ε, που διέπει όλη αυτή τη δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε στον Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αυτή, από αυτή τη σκοπιά τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη. Τελευταίο είμαι κύριε Πρόεδρε και θα σας δώσω το μικρόφωνο και το λόγο. Νομίζω ότι η τελευταία πρόκληση για τον νομοθέτη είναι η πρόκληση της ευθύνης, της υπευθυνότητας. Θα πρέπει δηλαδή να σχεδιάσουμε στρατηγικές, ε, αν θέλετε, αντιπαράθεσης με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν, ούτως ώστε ο χάρτης ε, να ε, έχει τη θέση που του αρμόζει και να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Είχαμε ε, επιτυχίες όπως με, το, τα στοιχεία PNR, με την οικογενειακή επανένωση. Θα πρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Και με το χάρτη των δικαιωμάτων. Και παραλαμβάνω, έχουμε την ευθύνη αυτή ε, που έχει ως στόχο να τηρήσουμε τις δεσμές που έχουν αναλάβει οι διάφοροι εκτελεστικοί οργανισμοί. Αυτό δεν αφορά την πολιτική εντολή, ε, αυτό αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους, αλλά πρέπει και κάθε εκτελεστικός οργανισμός να ε, τηρεί τις δεσμεύσεις του. Έχουμε λοιπόν μια επίπτωση που είναι σχετικά εύκολο να την καταλάβει κανείς και θα σας δώσω, θα μιλήσω για ένα λεπτό γι' αυτό. Μία από τι σημαντικότερε προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαδικασία για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ας το σκεφτούμε. Είπαμε ότι δεν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ των δύο κειμένων και αυτό θέτει σημαντικά προβλήματα. Δύο θα αναφέρω. Πρώτο στοιχείο. Η ρήτρα για την δημόσια τάξη Ξέρετε ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούσαν να αναφέρονται ε, ή να, να αντιμετωπίζονται από τον, τον δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε ένα θέμα αρμοδιότητας. Ε, στο δικαστήριο τυπικά η αναλογικότητα εξ ονόματος ε, της δημόσιας τάξης χαρακτηρίζει τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα μπούμε σε ένα σύστημα πραγματικά σχιζοφρενικό όπου θα πρέπει να αρνούμεθα ε, στους δικαστές μας ε, τη γνώση τέτοιων θεμάτων ενός άλλος δικαστής ε, εκτός από το Στρασβούργο δηλαδή θα μπορεί να τα πραγματεύεται αυτά τα θέματα. Πρώτο πρόβλημα. Και δεύτερο πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει έναν επικουρικό έλεγχο, δηλαδή μόνο όταν ε, δεν υπάρχει κανένα άλλο ένδικο μέσο ως δίκτυα ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα. Θα ολοκληρώσω λέγοντας το εξής κύριε Πρόεδρε. Η μελέτη του δικαίου σήμερα από πυραμιδικής και ιεραρχικής πλευράς ε, είναι παροχημένη πλέον. Φυσικά και υπάρχουν ιεραρχίες. Όπως όμως μιλάω για το κοινοτικό δίκαιο και λέω ότι η συνθήκη είναι πάνω-πάνω στην πυραμίδα, όταν μιλάω για το για δικονομικό δίκαιο ε, ή για οτιδήποτε άλλο, υπάρχει κορυφή της πυραμίδας και έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Η προσέγγιση που έχουμε σήμερα για το δίκαιο είναι πλουραλιστική και θα πρέπει να βάλουμε τάξη σε αυτόν τον πλουραλισμό. Και αν δείτε το πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων σήμερα, οι εθνικοί δικαστές, οι ανώτατα δικαιοδοτικά όργανα, τα συνταγματικά δικαστήρια των κρατών μελών, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιλαμβάνονται του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν και να τον κάνουν σεβαστό. Κανείς δεν σκέφτεται τι μπορεί να συμβεί αν ένας δικαστής στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία πάρει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ζητήσει την ερμηνεία του ή ερμηνεύσει μόνος του το χάρτη. Δεν μας απασχολεί αυτό. Πώς θα γίνει συνεργά, πώς θα υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ των δικαστών ώστε ο χάρτη να έχει αποτέλεσμα. Αυτό θα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ καθοριστικό. Και εν τέλει μήπως θα χρειαστεί να γίνει πλέον συνταγματική δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξελιχθεί δηλαδή και μέσω της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι με αυτό το τίμημα η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η... ο σεβασμός των αξιών της θα μπορέσει να εξασφαλιστεί. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μας είπατε πολλά και υπήρξατε πληρέστατο στην περιγραφή όλων των προκλήσεων που μας, που μας περιμένουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν πολλά ερωτήματα και απορίες. Δίνουμε λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Πριβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε σε αυτό το διακεκριμένο μέρος Επειδή όμως είμαι κρυωμένος μπορεί να μην εκφράζομαι πολύ σαφώς. Είναι βέβαια δύσκολο να μιλήσει κανείς μετά από τη διάλεξη του καθηγητού, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για τρία θέματα. Όπου υπάρχουν ελλείψεις στη χάρτα. Δεύτερον, τι άλλαξε από τότε που ενεκρίθη η χάρτα. Και τρίτον, ορισμένες συγκεκριμένες επιπτώσεις στον χώρο ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης. Το πρώτο σημείο όμως, ας το παραλείψω γιατί είπατε, ακούσατε ήδη πολλά για τη χάρτα, για να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Δεύτερο σημείο λοιπόν, τι έχει αλλάξει από τότε που ισχύει η χάρτα. Ακούσαμε και σήμερα και χθες ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε την χάρτα μέσα στα πλαίσια του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Αλλά αυτό δεν μας μαθαίνει τι, ποια ακριβώς είναι η φύση του. Επιτρέπει ασάφειες και παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. στο εξή τα εθνικά όργανα της Ένωσης και οι χώρες μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της χάρτας όποτε εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και άτομα και μη κυβερνητικέ οργανώσεις τώρα μπορούν να επικαλούνται τη χάρτα ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αυτό οδήγησε ορισμένα χάρη μέλη, κράτη-μέλη στην έκφραση φόβων ότι μπορεί να παραβιαστούν τα εθνικά του δικαστικά συστήματα. Παρά τους περιορισμούς του άρθρου 51.2 που λέει ότι η χάρτα δεν δημιουργεί καμία νέα δικαιοδοσία στην Ένωση παραδείγματος χάρη στην κοινωνική πολιτική, μπορεί και η απλή ύπαρξη ορισμένων τύπων δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο όπως τις ίσεις μεταχείρισης και της ισότητας γενικότερα να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα ιδιαίτερα αν μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο. Παρ' όλα αυτά δεν θα έπρεπε από αγωνιστικής απόψεως να θεωρήσουμε ότι η αντίσταση ή ο δισταγμός ορισμένων κρατών μελών στην πλήρη εφαρμογή μιας ε, δικαιοδοσίας ισονομίας σημαίνει ότι είναι απλά λόγια και δεν ε, ενδιαφέρεται κανείς στην πραγματικότητα για την όντως εφαρμογή τους. η χάρτα μιλά για ρητά δικαιώματα ισότητας και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό νομίζω ότι τα άρθρα 20 με 26 μπορούν να επικαλεστούν, μπορεί να, κανείς να τα επικαλεστεί κατά μια δημόσια αρχή ή κάποιο άλλο ατόμο. Επειδή όμω όλα αυτά περιορίζονται στι δικαιοδοσίε τη Ένωση και των κρατών μελών, δεν είναι σαφέ αν τα άτομα θα έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν αυτά τα δικαιώματα και αλλού. Είναι ενδιαφέρον ότι πρώτη απόψεως αυτά τα δικαιώματα εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα, σε όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτω εθνικότητα με την εξαίρεση του άρθρου 21.2 που απαγορεύει τη διάνυση μεταχείριση για λόγου εθνικότητα. Σύμφωνα με την συνθήκη τη Ένωση, αυτό εφαρμόζεται όμω μόνο στου πολίτε τη Ένωση και αποκλείει του τρίτου. Τα δικαιώματα που δημιουργεί η Χάρτα δεν είναι καινούρια, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα δεν είχαν συμπεριληφθεί στο κοινοτικό δίκαιο με τόσο ρητό και σαφή τρόπο ιδιαίτερα ως προς την ίση μεταχείριση με, για λόγους ε, εθνικούς ή φιλετικούς πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αναγνωριστεί ως θεμελιώδη δικαίωμα. Οι προβλέψεις της χάρτας λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ορισμένων δράσεων μη κυβερνητικών οργανώσεων για δράση κατά της άνησης μεταχείρισης και αντιρατσιστική δράση. Εκτός αυτού πρέπει να τονίσουμε ότι η χάρτα είναι πολύ προοδευτική στο εύρος και τη γλώσσα της διότι απαγορεύει οποιαδήποτε άνηση μεταχείριση με βάση τη φίλο, τη φιλή κτλ καθώς και οποιαδήποτε η μεταχείριση γενικότερα για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό σημαίνει ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό στο μέλλον και να το επικαλούνται. Τέλος, είναι χωριστά διατυπωμένο αυτό το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης και άρα δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Για πρώτη φορά γίνεται λόγος σε ενωσιακό κείμενο και για τα δικαιώματα μειονοτήτων. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η συμπεριφορά που επιφυλάσσουν στους τσιγκάνους, ιδιαίτερα στις καινούριε χώρες μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και τρίτον, τελευταίο, η επίπτωση της χάρτας σε ορισμένα συγκεκριμένα προγράμματα, επειδή έχει καθεστώς πρωτογενούς δικαίου η χάρτα, ο σεβασμός της είναι πια δεσμευτικός για, και για το δευτερογενές δίκαιο όπως τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Περιλαμβάνει ορισμένες ρήτρε που μπορεί κανείς να τις επικαλεστεί και ως προς πολιτική ασύλου και μετανάστευση. Παραδείγματος χάρη το άρθρο 19.2 απαγορεύει την έκδοση σε χώρα όπου ο εκδιδόμενος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο θανατικής ποινής βασανισμού ή άλλων απανθρώπων συμπεριφορών. Άλλα άρθρα μπορούν να αφορούν το δικαίωμα ή μη δικαίωμα κρατών μελών να επιβάλλουν περιορισμούς στα δικαιώματα των μεταναστών ή των συζύγων των. Όπως είπε και η Επίτροπος Ρέντινγκ, είναι σαφές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι βασική ρήτρα οποιασδήποτε νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Νομίζουμε ότι αν αυτό εφαρμοστεί στα σοβαρά και όχι απλώς στα λόγια, όπως έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές όπως ας πούμε για την ισότητα των φύλων, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό και να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών. Ως πρώτο συμπέρασμα λοιπόν νομίζουμε ότι η επίπτωση της χάρτας είναι ακόμη δύσκολο να αποτιμηθεί διότι θα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα την εφαρμόσουν τα το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Δικαστήρια. Αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όλο και περισσότερο γίνονται γνωστά τα δικαιώματα αυτά, ότι υπάρχουν δηλαδή και είναι γνωστό ότι όλη μια μέρα θα γεράσουμε, μπορεί να αρρωστήσουμε, μπορεί να αλλάξουμε φίλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό και πεπιθήσεις και μερικοί μπορεί να αλλάξουν και το χρώμα του θέρματός των. Γι' αυτό νομίζουμε ότι ο αγώνας για τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι αγώνας για ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας αλλά όλων των πολιτών. Όταν αυτό θα γίνει ευρύτερα γνωστό και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τότε ο χάρτης θα, έχει, θα αποκτήσει την πλήρη του σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν να προχωρήσουμε στους επόμενους δύο ομιλητές, βλέπω ότι κάποιος, ο κύριος Έντσιος ζητεί το λόγο. Θα συζητήσουμε λοιπόν λίγο τις δύο τελευταίες παρεμβάσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Λαβέ. Η παρέμβασή του δεν ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής αλλά κατάφερα να απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτηματικά που είχα εγώ. Εγώ προσωπικά και εκ μέρους των συναδέλφων μου θα ήθελα να σας παρακαλέσω και στο μέλλον να συνεργαστείτε στενότερα μαζί μου και αν είναι δυνατόν να μας δώσετε και γραπτός την παρέμβαση που κάνατε πριν από λίγο Ούτε ώστε να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν βάση και για μελλοντικέ μας εργασίες. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι τι είναι δυνατόν να προβλέψει κανείς τη χρονική στιγμή μέχρι την οποία αυτή η χάρτα των σεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Μπορεί κανεί να προβλέψει μέχρι πότε θα έχει γίνει αυτό και πιστεύετε ότι οι μηχανισμοί που φαίνεται να φαίνεται να φτιάχνονται. Πρέπει να είναι τέλειοι πριν να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα, διότι μια τελειοθυρία τέτοιου τύπου θα καθυστερούσε πολύ την υλοποίηση της χάρτας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, τη για τα σχόλιά σας αλλά ε, προσπαθώ να βρίσκομαι και μέσα στα χρονικά όρια τα οποία ορίζει ο πρόεδρος λοιπόν τώρα η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν τροποποιεί τίποτα σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Ένωσης και άρα δεν είναι υπονοεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα που ήδη τα κάνει σε τελευταία ανάλυση. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η σχετική ε, νομολογία είναι εφαρμόσιμη mm. έτσι, και από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη η χάρτα δεν επηρεάζει την κατάσταση αυτή. Όταν μιλάμε λοιπόν εδώ για τη χάρτα των συμμελιωδών δικαιωμάτων, μιλάμε για κάτι το οποίο ήδη υφίσταται, η δίκη, η δίκη, η απαγόρευση των διακρίσεων κτλ. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε. Ευτυχώς ζούμε σε δημοκρατικά καθεστώτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες αρχές ε, οι οποίες μπορούν να πηγαίνουν πολύ μακριά η καλή διακυβέρνηση, καλή διοικητική τάξη και τα λοιπά, η διαφάνεια και τα λοιπά. Αυτά είναι γενικότερα θέματα. Θα μπορούσα λοιπόν να σας πω, με ρωτάτε πότε θα εφαρμοστεί από όλους θεωρητικά μπορεί να εφαρμοστεί από όλους και αύριο γιατί είναι γνωστά τα πράγματα αυτά. Από την άλλη μεριά μπορώ να σας πω ότι δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί από όλους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επόμενο θέμα. Η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σχέση της με άλλα διεθνή μέσα και εργαλεία. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Η... Περιμέναμε πολύ καιρό και για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Και αυτό είναι λογικό βεβαίω, διότι από εκεί και πέρα υπάρχουν 27 κράτη-μέλη και αν το καθένα εφάρμοζε την ε, κοινωτική νομοθεσία όπω ήθελε, θα υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν όμω και άλλοι που όπως οι εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και τα λοιπά που δεν έχουν αποφανθεί και αυτό δημιουργεί μια κάποια ανισορροπία Απ' τη μια έχουμε την ομολογία κάποιων δικαστηρίων και απ' την άλλη έχουμε και κάποιους οι οποίοι ε, δεν έχουν ακόμη μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ακόμη πολλά πράγματα να σταθμίσει τα καλά και τα κακά πριν κάνει ένα επόμενο, επόμενο βήμα. Χτες ο δικαστής Μπονισό είπε ότι θα, το 10 ο Σονούπο θα εξέφραζε, θα έπαιρνε μία απόφαση πολύ σημαντική. Περί πρόκειται. Πρόκειται για κάτι αρκετά επίκαιρο στη Γαλλία ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Προδικαστικό ερώτημα που έφεσε γαλλικό εστιατήριο στο ΔΕΚ. Αλγερινοί συνελήφθησαν ε, στην Λίλα κατά τη διάρκεια ελέγχου ταυτοτήτων ε, κρατήθηκαν ε, για διοικητικούς λόγους το θέμα είναι αν πρέπει να απελευθερωθούν ή όχι. Δημιουργήσαμε λοιπόν πριν πάμε παραπέρα αν θέλετε στη Γαλλία ένα προδικαστικό ερώτημα ε, προς το ΔΕΚ ε, για να δούμε τι έχει να πει η Ευρώπη, το, διοικητικό, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και βεβαίως ε, υπάρχουν και αντιρρήσει στη Γαλλία για αυτή τη δικαστική διαδικασία αλλά τέλος πάντων το ΔΕΚ λέει ότι το εφετείο στη Γαλλία το οποίο με τη διαβίβαση αν θέλει και το προδικαστικό ερώτημα έχει δίκιο στο να λέει ότι θα πρέπει να αποφασίσει πρώτα το ΔΕΚ για αυτό το θέμα. Άρα η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή ε, είναι αντικείμενο και αρμοδιότητα αν θέλετε των εθνικών δικαστηρίων και οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται σε πρώτη φάση εκεί και τώρα. Με... Υπήρχε αυτό πιο πριν, θα μου πείτε, ωραία, για κάποια τέτοια θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τώρα με τη χάρτα ε, ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Και βεβαίως υπάρχουν προκλήσεις, αλλά άμα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, ε, μόνο τότε θα μπορέσει να φτιαχτεί μια Ευρώπη που να ανταποκρίνεται σε αυτό που προσδοκούν, που θέλουν οι πολίτες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Α, παρακαλώ. Παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που ξύπνησα λίγο αργά τελικά στη συζήτηση. Καθυστέρησα να έλθω κιόλος και δεν κατάφερα να, ακούω, να ακούσω όλη σας την παρέμβαση. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαι ο παδός όμως της χάρτας γιατί πιστεύω ότι έτσι υποβασμίζεται, αν θέλετε η σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αλήθεια αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι ή πώς βλέπετε το μέλλον σε δικαστικό επίπεδο και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί και τι αρμοδιότητε. Euh, Είναι ένα λεπτό θέμα, ε, θα, δεν θα ήθελα ε, να το σχολιάσω, θα μπορούσα τέλος πάντων να επεκφύγω, αλλά παρόλα αυτά. Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά διδάγματα που μας ε, έδωσε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και που θα τεθεί και με τη χάρτα, με το χάρτη, είναι η ιδέα σύμφωνα με την οποία η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν σταματά εντός των συνόρων. Η εξοεδαφική ισχύς εμβέλεια των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτεί στις σχέσεις που μπορούμε να έχουμε με τρίτες χώρες οι αξίες που σεβόμαστε καθ' ολοκλήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλλονται με την ίδια ισχύ. Και αυτό ακριβώς είναι, αυτή ακριβώς είναι όλη η συζήτηση και το θέμα με το SWIFT. Και σε αυτό το τομέα δεν θα τολμήσω βέβαια, επαναλαμβάνω, να μπω σε ευαίσθητο έδαφος ε, υπάρχουν οι σημαντικές ευθύνες που υπάρχουν. Είναι άλλοι φορείς που και άλλα θεσμικά που ενδεχομένω να μην έχουν τόσο πολύ μεγάλη ευαισθησία για τις υποχρεώσεις τους. Όμως, δεν χρειάζεται να κατηγορούμε ή να υποπτευόμαστε για κακή πρόθεση τους εταίρους μας συστηματικά. Αλλά υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, μια συνειδητοποίηση και νομίζω ότι αυτό έχει καταστροφική επίπτωση ε, σε πρακτικές και μεθόδους που γνωρίζαμε παλαιότερα. Είμαστε περήφανοι και εδώ ακόμη ε, για τις πτήσεις της ε, CIA που τελικά συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας είτε σε επίπεδο κρατών μελών είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκε να δείξει με το δάκτυλο Dick Μάρτι τι... και να πει τι συνέβη. Πραγματικά βρισκόμαστε ε, σε μία δίνη κατά κάποιο τρόπο. Ε, νομίζω ότι δεν το συνειδητοποιούμε ακριβώ. Χάρη ε, στην επίπτωση που έχει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, προ το παρόν έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μόνο, αλλά μετά θα έχουμε και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και ίσως να χρειαστεί να ακολουθήσουμε δύο αντίθετε μεταξύ του κατευθύνσεις. Έχουμε και κάποια αντιδημοκρατική νομοθεσία μετά, το, μετά τα γεγονότα του Λονδίνου. Υπήρξε η νομοθεσία αυτή, καταδικάστηκε από τη Βουλή των Λόρδων. Και υπήρξε μια σχετική υπόθεση, η οποία πήγε στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά απόλαυσα κάθε λέξη τη απόφασης ε, και πρέπει να σας πω ότι η απόφαση αυτή, το δικαστήριο αλλά με πολύ υποκριτική διάθεση ε, και προσποιούμε εντελώ, λέω ότι πραγματικά εκπλήσωμαι. Δεν έχω ξαναδεί ε, να επικρίνει ουσιαστικά ε, τους εθνικούς του δικαστές μια χώρα ενώπιόν λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει στο, Ευρωπαϊκό, στο Ενωμένο Βασίλειο βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καλεί στην τάξη τους ε, εθνικούς δικαστές, τους βρετανικούς δικαστές. Επομένως, ο κόσμος του χθες έχει πεθάνει, βρισκόμαστε σε ένα νέο κόσμο όπου οι δικαιοδοσίε και οι νομοθέτες θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμβατές ερμηνείες. Δεν μίλησα για την εξοδικαστική ισχύ, το εξοδικαστικό αποτέλεσμα εξοεδαφικό αποτέλεσμα. Έχουμε κάποιες άλλες, ε, κάποια άλλα παραδείγματα ε, της ειρηνευτικές διαδικασίες, ε, μίλησα για μετανάστες που μπορεί να βρεθούν σε διεθνή ύδατα μέσα σε μια σχεδία κτλ. Εμείς, εμείς σε εμάς εναπόκειται, μάλλον σε εσά θα έλεγα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναπόκειται να φροντίσετε ώστε αυτό τα οποία θα γίνονται από την άλλη πλευρά θα είναι ε, στο ύψος αυτό που θα μπορούσαν να εσωτερική αγορά, ε, τα νομισματικά οικονομικά θέματα. Αυτές είναι οι προκλήσεις. Και νομίζω ότι ο χάρτης είναι ένα αυτόνομο εργαλείο το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εξασφαλιστεί εδώ. Και κανεί δεν θα πρέπει να κρύβεται πίσω από το μικρό δάχτυλο. Merci. Euh, Βλέπω ότι δεν θέλει κάποιος να παρέμβει, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την για διάταξη και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ήμον Μακάουντα, που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας ε, των Εθνικών Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας Χαίρομαι ακόμη πιο πολύ γιατί μας καλέσατε να είμαστε εδώ εκ μέρους όλων των εθνικών ε, θεσμικών οργάνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η, τα θεσμικά αυτά όργανα είναι εθνικά, είναι ανεξάρτητα από την κοινωνία και βρίσκονται σε ένα σε μια τρίτη διάσταση αν θέλετε και η, ομάδα αυτών των ε, θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκή Ομάδα που δημιουργήθηκε το 2006, εκπροσωπεί 34 περίπου, 34 θεσμικά όργανα από ολόκληρη την Ευρώπη, 20 εκ των οποίων έχουν επιστοποιήσει με βαθμό α σύμφωνα με τις αρχές των ε, Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές του Παρισιού όπως λέμε. Είναι πολύ σημαντική ομάδα αυτή λοιπόν θεσμικών οργάνων που ε, προσπαθεί να συνδυάσει τα διεθνή πρότυπα ε, και τους ελέγχους που γίνονται ε, από το διεθνές σύστημα, σύστημα με τα αντίστοιχα των εθνικών συστημάτων. Ε, καν έχουμε η ομάδα αυτή έχει πολλά πολλές αρμοδιότητες και δρά ε, και σε σχέση με τα δικαστήρια και σε σχέση με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και ε, έχει στενές σχέσεις και με τον οργανισμό, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου ο οποίος οργανισμός αναγνωρίζει το ρόλο των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Α, αναφέρεται στο καταστατικό, στο ιδρυτικό κανονισμό μάλλον της του οργανισμού της Βιέννης ε, ότι είναι απαραίτητη σχέση με τα εθνικά θεσμικά όργανα. Στην ε, ε, τελευταία μας μελέτη, στην τελευταία μας έρευνα που κάναμε που έκανε μάλλον ο οργανισμός της Βιέννης υποστήριξε τη δημιουργία και ενίσχυση αυτών των εθνικών θεσμικών οργάνων σε όλα τα κράτη-μέλη. Μοναχά δεκα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν τέτοιου είδους θεσμικά όργανα που συμμορφώνονται πλήρως μετά. Ε, με τις αρχές του Παρισιού. Έξι ακόμη κράτη-μέλη ε, έχουν τέτοια όργανα τα οποία δεν συμμορφούνται πλήρως με τις αρχές του Παρισιού και επιπλέον ο οργανισμός της Βιέννης σύστησε να υποστηρίζονται τα εθνικά θεσμικά όργανα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συνεργάζονται και διεθνώς. Υποστηρίζουμε τις συστάσεις αυτές της φρά και πραγματικά ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους δεσμούς αυτούς. Τώρα ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ρόλοι, ο ρόλος που έχουν να παίξουν τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η, η χάρτα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βοηθήσει πέρα από ορισμένα πράγματα που τα γνωρίζουμε ως θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και στην ε, ανάπτυξη της έννοιας της ευρωπαϊκής ε, να δημιουργήσει μια, ένα χώρο ε, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης να ενισχύσει την ε, νομική βεβαιότητα όλων των πολιτών της Ένωσης βεβαίως υπήρχε τέτοια προστασία και στο παρελθόν αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν όλες αυτές οι έννοιες για τον πολίτη ούτως ώστε ο πολίτης πραγματικά να μπορεί να κατανοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρά και σε εθνικό επίπεδο και τη συσχέτισή του με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να δουλέψουμε για να τονίσουμε και να εξασφαλίσουμε στο μέλλον τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, βρίσκονται στο πυρήνα οποιασδήποτε νομοθετικής πρωτοβουλίας παίρνετε, οποιασδήποτε χάραξης πολιτικής, είτε πρόκειται για άσυλο, είτε πρόκειται για λαθρεμπόριο ατόμων, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, θα πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα των ευρωπαϊκών, ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πραγματικά η καθημερινότητα των πολιτών της Ευρώπης συνδέεται με τα θέματα αυτά, δεν είναι απόμακρα. Η... Πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα προσφύγων, τουν τον άσυλο στα διάφορα σύνορα, ε, σωματεμπορίου, απελαθρεμπορίου, ανθρώπινων όντων κτλ δεν θα πρέπει να τα αγνοούμε λοιπόν για να μην υποτιμούμε τη, δυνα... τη σημασία της ε, πραγματικής υλοποίησης της ε, Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τελειώντας θα ήθελα να πω πόσο χαίρομαι που η κυρία η Επίτροπος Vivian Redding ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο τα θέματα της ε, αυτά και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομάδας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ιρλανδίας θα συναντηθώ με την Επίτροπο την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 για να μπορέσουμε να οργανώσουμε με πιο συγκεκριμένη και στενή συνεργασία. Σας υπόσχομαι ότι υπό την ιδιότητά μου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Εθνικών Οργανισμών και εκ μέρους της ε, Ιρλανδίας αγωνιστώ μέχρι ε, τελευταία δρανίδος για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο David Nichols, Διεθνής Αμνηστία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να επανέλθουμε στο πώς ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατ' επέκταση η ολόκληρη κοινωνία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χάρτα για να και κατά ορισμένων αρχών. Καταρχήν μερικά γενικά θέματα που σκεφτόμαστε όταν βλέπουμε τη χάρτα όσα έχει τώρα. Πρώτον, είναι το πρώτο κείμενο από τότε που ο ΙΕ ίδρυσε την υπάτη αρμοστία που αναφέρει πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα μαζί. Και είναι τεράστια η σημασία του για μας στην Διεθνή Αμνηστία και γενικότερα για το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί συνεισφέρει στην επίγνωση του αδιέρετου χαρακτήρα των δικαιωμάτων αυτών όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά και στην εξωτερική της πολιτική. Δεύτερον, διαφωνώ λιγάκι με αυτά που είπε ο καθηγητής Λαμπέλ. Δηλαδή εμείς δεν θεωρούμε το, τη χάρτα ως ιδιαίτερα επαναστατική. Για μας το κυριότερο είναι ότι επαναβεβαιώνει τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει και συνυπογράψει η Ένωση και διεθνώς. Εδώ θέλω να συμφωνήσω με τον άλλο μιλητή που μίλησε για το συνδυασμό της με, τη διεθνή, με το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε να αναφέρουμε τη χάρτα αλλά και τις ρήτρε του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν περιγράφουμε τη σημασία της χάρτας σε άλλες χώρες για τις οποίες θα είναι λιγότερο σημαντική η χάρτα. Για να μην θεωρηθεί ότι η Ένωση επιβάλλει τα δικά της, τις δικές της αρχές σε άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, η χάρτα περιλαμβάνει νέα δικαιώματα. Ήδη μιλήσαμε για το άρθρο 8 προστασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει και το 41 που μιλάει για την καλή διακυβέρνηση ή καλή διαχείριση πράγμα το οποίο δίνει νέες δυνατότητες στην κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης έχει νέες διατυπώσεις. Το είπε αυτό ο καθηγητής Λαμπέλ. Ως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα το 21 για την ίση μεταχείριση, αλλά και το 9 για τους γάμους. Όπου αντίθετα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ο γάμος δεν περιορίζεται μόνο σε αντίθετα φύλλα. Επίσης ε, αποσαφηνίζει ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν παραλυφθεί ή δεν αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο, όπως το 19.2. Το 19.2. Τρίτο γενικό θέμα που θέλω να θίξω. Είναι πολύ σημαντικό ότι η χάρτα δεν εφαρμόζεται μόνο στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά σε όλους όσους υπόκεινται στον Ευρωπαϊκό νόμο. Μάλιστα ο τίτλος του αναφέρεται συγκεκριμένα σε δικαιώματα των πολιτών, αλλά δεν εννοεί μόνο τους ε, πολίτες της Ένωσης. Το 41, 42 και 45 2 αφορούν και όλους όσους ζουν στην ενωσιακή επικράτεια και στους οποίους εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Τέλος, υπάρχουν ακόμη πολλές ασάφειες στη χάρτα που πρέπει να αποσαφινιστούν μέσω της, ε, των περιπτώσεων που θα εκδικαστούν περίπτωση την περίπτωση με την ομολογία δηλαδή παραδείγματος χάρη η χάρτα είναι ασαφής ως προς το διαχωρισμό μεταξύ αρχών και δικαιωμάτων. Αυτό εξηγείται λίγο περισσότερο στο συνοδευτικό κείμενο, αλλά όχι στο κυρίως. Πρέπει αυτό να δοκιμαστεί μέσω συγκεκριμένων περιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και από το Κοινοβούλιο. Τώρα, πιο πρακτικά, πώς ακριβώς θα μπορούσε η κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τη χάρτα. Είναι σαφές ότι σε δύο μέτωπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το πρώτο είναι να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία και όλες οι προτάσεις της Κομισιόν εφόσον περνούν από το Κοινοβούλιο θα διορθώνονται ώστε να συμφωνούν πλήρως με τη χάρτα. Και δεύτερον το Κοινοβούλιο και η Κοινωνία των Πολιτών θα μπορούν να την επικαλούνται έναντι άλλων θεσμικών οργάνων. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τρεις τομείς. Ένα για την αντιτρομοκρατία που το αναφέραν και προηγούμενοι. Δεύτερον για την ίση μεταχείριση και τρίτον για θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Για την αντιτρομοκρατία Οι διατάξεις της χάρτας δίνουν στο Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών πιο σαφείς ιδέες ως προς το πώς πρέπει οι προτάσεις της Κομισιόν αλλά και η δράση των άλλων θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών να συμμορφώνονται στο μέλλον. Παράδειγμα, η μαύρη κατάλογη υπόπτων τρομοκρατίας πριν γίνει νομικά δεσμευτική η χάρτα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε ήδη αποφασίσει ότι πρέπει να πληροφορείται κάποιος αν έχει εγγραφεί σε μαύρο κατάλογο. However, this is, this is still not in with... Και αυτό θα συμφωνούσε και με το διεθνές δίκαιο. Είναι θέμα πρόσβασης σε δίκαια δίκαια αλλά και θέμα καλής διαχείρισης. Το σχετικό άρθρο λέει ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων αν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση εις βάρος του. Πολλές από τις χειρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είδαμε τα τελευταία χρόνια ως προς την αντιτρομοκρατία δεν καθορίζονται σαφώς μεταξύ των δικαιοδοσιών της ΚΕΠΑ και της υπόλοιπης Ένωσης. Συχνά λέγεται ότι η χάρτα δεν καλύπτει την ΚΕΠΑ. Δεν αφορά την εξωτερική πολιτική. Δεν είναι σαφές αυτό. Το είπαν και άλλοι. Η χάρτα είναι δεσμευτική για όλα τα θεσμικά όργανα και σώματα της Ένωσης τα οποία πρέπει να σέβονται τη χάρτα σε όλες τους τις πράξεις. Το Συμβούλιο και την Προεδρία του, το Frontex και άλλα ιδρύματα, καθώς και την εξωτερική υπηρεσία και την αντιπροεδρία της Κομισιόν. Εφόσον είναι λοιπόν δεσμευτική για όλα αυτά η χάρτα, τότε έπεται ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ίδιο δεν έχει δικαιοδοσία για την ΚΕΠΑ. Παρόλα αυτά είναι υπόλογα τα όργανα αυτά ως προς το δικαστήριο για να σέβονται τη χάρτα, ως προς το σεβασμό της χάρτας. Και αυτό θα δοκιμαστεί τα επόμενα χρόνια. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη επικαλεστεί τη χάρτα κατά τις διαπραγματεύσεις SWIFT. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και για άλλες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Παραδείγματος χάρη για την αμοιβαία νομική υποστήριξη και τις εκδόσεις. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για την συμμεταχείριση, έχουν καλυφθεί από άλλους. Θα ήθελα απλώ να πω ότι σημαντικό μέρος της χάρτας αφορά το θέμα ακριβώς αυτό και προσθέτει καινούργια επιχειρήματα όπως τον σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες διακηρύξεις. Επίσης τα δικαιώματα των τσιγκάνων και το, το δικαίωμα του εκλέγες θέτων. Τέλος για την άσυλο και, το άσυλο και τη μετανάστευση. Ανέφερα ήδη το 19.2 για πρώτη φορά αναφέρει ρητά ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ζωτική. Και δεν αφορά αυτό μόνο όσου ζητούν άσυλο, αλλά και εκείνου που μπορεί να εκδιωχθούν για επιστροφή, για να έκδοση δηλαδή, για να αντιμετωπίζουν απειλή θανατικής καταδίκης κλπ. Σήμερα αυτό απαγορεύεται ρητά και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει η κοινωνία των πολιτών και άλλοι, καθώς και άλλες. Το 41 για την καλή διαχείριση. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι ελλείψεις της δημόσιας διοίκησης ζημιώνουν πολύ κόσμο παραδείγματος χάρη για την ανανέωση εγγράφων ή, ή ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή θεμάτων επανένωσης οικογενειών. Τώρα θα μπορεί κανείς να επικαλεστεί το άρθρο αυτό στα εθνικά δικαστήρια. Τέλος, για το άρθρο 1, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το άρθρο 1 θεωρεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως την απόλυτη βάση της χάρτας. Και αυτό φυσικά είναι σημαντικό όταν ε, βλέπει κανείς θέματα ασύλου και μετανάστευσης ιδιαίτερα. Επίσης έχει τεράστια σημασία για τη δική μας της Διεθνούς Αμνηστίας καμπάνια για την αξιοπρέπεια και για τον τονισμό του αδιέρετου χαρακτήρα όλων των δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε κύριε Νίκος. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για συζήτηση. Αν κανείς ή καμία θέλει να θέσει κάτι, ορίστε εσείς εκεί κάτω ποιος είστε. Έχετε το λόγο. Τζαν Μικέλη Τζορτάνο λέγομαι. Είμαι Ιταλός και είμαι αρμόδιος για τις διαβουλεύσεις για τα ευρωπαϊκά θέματα στις Βρυξέλλες. Λυπούμε που δεν ήμουν παρόν από την αρχή στη συζήτηση. Αλλά αν μου επιτρέπετε να κάνω τα ερωτήματά μου στα Ιταλικά. Το πρώτο ερώτημα αφορά το δικαίωμα ασύλου πριν από λίγο καιρό νομοθέτησε η χώρα μου συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά ε, κάποιους μετανάστες τους οποίους ε, ε, βρίσκαμε στα διεθνή ύδατα. Υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις και ο επατσαρμοστής του ΙΕ αντέδρασε και η κυρία Ρέντινγκ. Πρώτο ερώτημα λοιπόν, τι μπορούμε να συναγάγουμε αυτή τη στιγμή όταν πολλά ε, είναι αντίθετα με τις διατάξεις ευρωπαϊκές. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ε, ιδιωτική ζωή. Στην Ιταλία γίνεται λόγος για μια πρόταση νόμου που θα έχει ως στόχο την απαγόρευση δημοσίευσης ε, των, του προϊόντος τηλεφωνικών υποκλοπών στις εφημερίδες. Και υπάρχει εδώ ένα θέμα ασυμβατότητας ή σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα. Δεν ξέρω. Ίσως θα μπορούσαμε να μας πούν οι ομιλητές σας κάποια θε... να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Άλλοι θέλουν το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ από το Euroline. Είμαι μια μη καπαόμικρον που εργάζεται για τις ε, γλωσσικές μειονότητες στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες, ε, για κάποιες καταστάσεις που έχουμε ε, στη Βρετάνη. Σλοβακική, Ουγγρική, γλωσσική μειονότητα. Τι γίνεται όταν κάποια κράτη-μέλη απέχουν τόσο πολύ από τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά τη μη διάκριση για λόγους γλώσσας. Παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τεράστια βήματα, αλλά κάποια κράτη-μέλη δεν ακολουθούν από ό,τι φαίνεται σε ό,τι αφορά την ισότιμη μεταχείριση. Ακούσαμε την Επίτροπο να λέει σήμερα το πρωί ότι με την εσωτερική πολιτική των χωρών για τις γλώσσες δεν μπορεί κανείς να παρέμβει. Πώς θα γίνει η συμφιλίωση αυτή. Βοηθούμε να υπάρχει μια αποσύνδεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο. Δεν βλέπω να σηκώνεται κανένα χέρι. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Ας επανέλθω λοιπόν στο πάνελ. Φαντάζομαι ότι ο καθηγητής Ροντοτά, γιατί σε αυτόν και ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ίσως θα ήθελε να το σχολιάσει. Θα μπορούσατε ίσως για την Ιταλική κατάσταση να μας τα πείτε εσείς καλύτερα και μετά θα ακούσουμε τους ε, εκδεξιών μου πανελίστες για τα υπόλοιπα θέματα. Καθηγητέ Ροντοτά, θα θέλατε το λόγο. Σε ό,τι αφορά τα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία και έχουν σχέση με τη χαρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι έμεσα διασαφηνίστηκαν με μία δήλωση που έκανε πριν από δύο ημέρες η κυρία Ρέντινγκ, την οποία είχαμε τη χαρά να ακούσουμε και σήμερα το πρωί. Η κυρία Ρέντινγκ στη δήλωσή της υπενθύμησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με τα προσοχής την κοινοβουλευτική διαδρομή αυτού του νόμου, του Ιταλικού, και θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το άρθρο 11. Δηλαδή, το άνθρωπο που αφορά την ελευθερία έκφρασης ε, και την ενημέρωση. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αντλεί από, την, από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιών. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό τον νόμο. Άλλωστε δημοσία και επανειλημμένο στην Ιταλία τον έχω επικρίνει. Δεν είμαι εδώ όμως γι' αυτό. χθες η συζήτηση ε, κάλυψε και κάποια άλλα θέματα πιο γενικά τα οποία καλύπτονται και από το χάρτη και συγκεκριμένα Τι μέλη με την ε, προστασία των ε, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι λίγο διαφορετική, ε, διαφορετική από την, μάλλον από την ιδιωτική ζωή, τη προστασία της ιδιωτικής ζωής, που ήταν λίγο διαφορετικά διατυπωμένη ως αρχή στο άρθρο 7 ήταν αρχικά και μετά προσθέθηκε ένα άρθρο 8 ειδικό για την προστασία των δεδομένων η σχέση μεταξύ της νέας διάστασης προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος ε, στην ενημέρωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη δύο πράγματα, δύο στοιχεία. Που νομίζω ότι είναι εμφανή και στον ίδιο το χάρτη. Από αφενός δηλαδή υπάρχει το δικαίωμα στην ενημέρωση, αλλά και η ανάγκη ισορροπίας εξισορρόπησης των διαφόρων συμφερόντων. σε σχέση με θεμελιώδη ζητήματα που αναφέρονται στη χάρτα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το άρθρο για την καλή διαχείριση και για τη διοικητική διαφάνεια που λαμβάνει υπόψη η χάρτα. Αν το δούμε, συνειδητοποιούμε ότι η ελευθερία έκφρασης ενισχύεται κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία προστασία των άλλων αξιών, δηλαδή χρηστή διαχείριση, ουσιαστικά καλή διεξαγωγή της πολιτικής δραστηριότητα. Και υπάρχει μια άλλη αρχή η οποία προέρχεται κυρίω από τη ΣΥΠΑ αλλά ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία κατοχυρώνεται με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι για δημόσια πρόσωπα, για πολιτικούς που έχουν σημαντικά αξιώματα δημόσια υπάρχει δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας και αυτό υπερέχει του ε, δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Όχι ότι εγκαταλείπεται το δικαίωμα αυτό, απλά ε, υπερτερεί γενικότερη αυτή η θεώρηση. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Δηλαδή, και επανέρχομαι με αυτό σε κάτι το οποίο ανέφερα στην παρέμβασή μου και το οποίο ανέφερε και ο καθηγητής Λαμπέλ. Ουσιαστικά πρόκειται για το εξής. ως νομικά ε, δεσμευτικό έγγραφο αυτή η χάρτα αυτά τα χρόνια ακόμη και αν δεν είχε την πραγματική νομική ισχύ μιας συνθήκης αναφέρεται σε πάμπολες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά και από πολλά εθνικά ε, δικαιοδοτικά όργανα. Και αυτό το αναφέρω γιατί υπάρχει πραγματικά ένα κεκτημένο, υπάρχει μια κληρονομιά. Και ίσως θα ήταν χρήψιμο να σκεφτούμε όλα αυτά. Η νομολογία κατά κάποιο τρόπο έχει τονίσει και μια κριτική που είχε, ε, ότι μια κριτική, η κριτική που είχε γίνει για, τη, για την χάρτα ήταν αδικαιολόγητη, ήταν αβάσιμη. γιατί πρόκειται ουσιαστικά για μια άλλη έκφανση της οικονομίστικης ε, ε, θεώρησης. Όχι, εδώ έχουμε μη με την ε, λογική αυτή και το βλέπουμε και στο κείμενο της χάρτας. Η νομολογία και αυτές οι εκατοντάδες των αποφάσεων ουσιαστικά μας δείχνουν ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο έχοντας ως γνώμονα ε, τη χάρτα. με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, που μπορεί να έχονται σε αντίθεση με, τα, με τις ε, επιταγές της αγοράς. Υπάρχει στην Ιταλία και το λέω υπόψη της Επιτροπής ε, μία στοσελίδα ε, η οποία δημιουργήθηκε με συνεργασία των ε, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών διαφόρων κρατών μελών. Μπορούν να βρουν εκεί αποφάσεις διάφορες γλώσσες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Το λέω και για να σας δώσω μια επιπλέον πληροφορία αλλά και για να παρατηρήσω και να, επιβεβαι... να ε, τονίσω αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι ναι μεν τα δικαστήρια είναι ιδιαίτερα ενεργά και δραστήρια και ήταν και είναι και θα είναι, σήμερα υπάρχει επιπλέον η ιδιαίτερη ευθύνη για το νομοθέτη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλιώς την Ευρώπη θα την κάνουν οι δικαστές. έχει ξεκινήσει διαδικασία αναγνώρισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που σήμερα καταλήγει με αυτή τη χάρη. Ευχαριστώ. Πριν ε, πουν ε, οι δεξι, εκ δεξιών μου την άποψή του, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τζάρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο λόγια μοναχά για το άσυλο. Στις αρχές του φθινοπόρου ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της, Βιέννης, της Βιέννης θα έχει κάποιες μελέτες μάλλον θα ξεκινήσει κάποιες μελέτες ε, στα διάφορα κράτη-μέλη, στα διάφορα σύνορα ε, προς να δει ακριβώ ποια είναι η κατάσταση επιτόπου. Ελπίζουμε ότι η πρώτη έξεση θα είναι έτοιμη γρήγορα και θα σχετίζεται με την κράτηση στα σύνορα. Τώρα, επανέρχομαι σε ένα από τα προηγούμενα θέματα, όπου ε, δεν εφαρμόζουμε... Όντως, πρώτη δεν εφαρμόζουμε μόνο τα ε, ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και αυτά των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Όταν παραδείγμα παραδείγματο χάνει και θα το δείτε στη μελέτη ε, αξιολογούμε την κράτηση στα σύνορα. Ήρθαμε σε επαφή με 300-400 άτομα ανήλικους σε 5-6 χρόνια για να δούμε και τι ε, Προβλήματα υπάρχουν. Αυτή είναι η δεύτερη μελέτη που ενδιαφέρει για τους ανήλικους στα σύνορα. Τρίτη η μελέτη θα σχετίζεται με την νομική αρρωγή που παρέχεται σε αυτούς τους ε, μετανάστες τι είδους ε, διαδικασίες υπάρχουν κατά πόσον όλα αυτά είναι συμβατά και συμμορφούνται με τα πρότυπα ε, αυτά όλα είναι σοβαρότατα θέματα και κάπου συνδυάζονται αν θέλετε και με τις συζητήσεις που γίνονται στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Τζάραμπ. Thank you. Ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το θέμα του ασύλου βεβαίως οι συνάδελφοί μας από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι για να κάνουν έναν πλήρη αν θέλετε κατάλογο των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν αλλά θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι εν πολλοίς υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής που υπευλήφθησαν από την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βελτιώσεις ε, που απαιτούνται στην ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και ότι πρέπει να, να επιδιωχθεί αν θέλετε μια κάποια εναρμόνιση προς τα πάνω να εξασφαλιστεί ότι η οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα α, τηρούνται, γίνονται σεβαστά. Και βεβαίως μιλούμε για την ανάγκη όλα αυτά να εφαρμόζονται σε όλους. Ε. Τώρα, για την ε, Ιταλία. Θα ήθελα να πω ότι ο είπα αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα επισκέφθηκε την ε, Ιταλία το Φεβρουάριο που μας πέρασε και όντως τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της μετανάστευσης και του ασύλου είτε είχαν ε, υψηλή προτεραιότητα. Δεν ε, θα προσπαθήσω τώρα να απαριθμίσω όλα τα προβλήματα εφόσον δεν έχουμε και πολύ χρόνο και φόσον και η επίσκεψη διήρκεσε μόνο δύο μέρες. Ωστόσο έγιναν πολλές επισκέψεις και στα στην κυβέρνηση, σε μέλη της κυβέρνησης και στο, στην κάτω και στην άνω βουλή και είδαμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία εκεί. Παραδείγματος χάρη ο αριθμός των ασύλων που, του των ατόμων που στα οποία παρέχεται άσυλο, είναι αρκετά υψηλός. Υπάρχουν όμως βεβαίως και προβλήματα όπως η όλη πολιτική ένταξη ε, σε συνδυασμό με την ασφάλεια ε, τα κλισέ τα στερεότυπα των μαζικών μέσων ενημέρωσης που συνδέουν τους ε, αλλοδαπούς με την εγκληματικότητα και προβλήματα υπάρχουν και την εθνική πολιτική το που φαίνεται να είναι εθνική πολιτική ε, αν θέλετε προς την Λιβύη των σκαφών που, που περιέχουν μετανάστες. Εκεί παίζει και η σύμβαση της Γενέβης βεβαίως. Και Βεβαίω η δικαιολογία που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν η Ιταλία ήταν ότι οι, τα Ηνωμένα Έθνη δεν συναλλάσσονται με τη Λιβύη. Αυτό όμω ίσχυε στο παρελθόν, δεν ισχύει απαραίτητο τώρα. Αυτό το είπε πάντως ο είπα αρμοστής, είπε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, είναι ένα παράδειγμα ρεφουλμό όπως λέμε, ενώ βίαιου επαναπατρισμού τελικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζάρα, προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια, το δεύτερο μιλητή ο κύριος και μετά θα πάρετε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ με τα προβλήματα των κυρίων από το Eurolang. Υπάρχει μία σύγχυση ως προς το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Και αυτό δεν βοηθιέται καθόλου από το ότι έχουμε αντιφατικά μηνύματα από τα διάφορα όργανα εδώ αλλά και από τα, τις χώρες μέλη ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Το μόνο που μπορώ να σας πω για να σας παρηγορήσω είναι ότι πρώτα πρέπει να δούμε μήπως αποσαφινιστούν αυτά τα πράγματα στην, στην επόμενη δήλωση της Επιτροπής αλλά και πριν από αυτό δεν είναι θέμα αποκλειστικά των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον η χάρτα, αλλά, αλλά και των πολιτικών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις Εθνικές Βουλές. Οι εθνικοί βουλευτές πρέπει να γνωστοποιήσουν τα προβλήματα αυτά στις κυβερνήσεις τους και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ήδη ότι αυτό που ακούγεται είναι μαξιμαλιστική προσέγγιση ως προς την χάρτα. Το Κοινοβούλιο δηλαδή δεν θα περιμένει τον Οκτώβριο, αλλά ήδη από τώρα θα χρησιμοποιήσει τη χάρτα, τη χρησιμοποιεί και τις παραπομπές στο Διεθνές Δίκαιο για να τροποποιήσει και να διορθώσει την νομοθεσία και καλεί από τώρα και τα άλλα όργανα και για θέματα εξωτερικής πολιτικής να τη διορθώσουν. Ο κύριος Μακόντα. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Καταρχήν, φυσικά και εμείς ελπίζουμε η επόμενη δήλωση της Κομισιόν να είναι πιο σαφής. Δεύτερον, τη σημασία που έχουν οι εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο για το άσυλο και τη μετανάστευση που εκφράζονται στην πράξη εθνικά αλλά και ως προς την διατύπωση γενικότερων προτύπων πανενοσιακά που στόχος τους είναι να λειτουργήσουν καλύτερα οι εθνικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πρίβος. Η χάρτα δεν είναι μεν εφαρμόσιμη παρά μόνο για θέματα ενωσιακής δικαιοδοσίας και στα κράτη-μέλη, αλλά ως μη κυβερνητική οργάνωση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο και δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ενημέρωση της νομοθεσίας για να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για τη χάρτα. Είναι λοιπόν χρήσιμο να αρχίσουμε να κάνουμε ένα είδος monitoring χρησιμοποιώντας τις διατυπώσεις της χάρτας όπως το 21 ως μήκη όμικρον ακόμη και αν τα θεσμικά όργανα καθυστερήσουν. Ευχαριστούμε κύριε Πριβό. Καθηγητής Λαμπέλ θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ. Μόνον ότι όλα αυτά είναι πολύπλοκα διότι εάν τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελέσουν ένα είδος κοινού παρονομαστού το παρόλα αυτά έχει ο καθένας και τις δικές του νομικές παραδόσεις και ιστορικό παρελθόν και είναι γι' αυτό μεγάλη πρόκληση σήμερα στην Ένωση το πώς θα κατορθώσουμε να εξισορροπήσουμε, πράγμα που είναι απαραίτητο, όλες αυτές τις διαφορετικές παραδόσεις, ώστε να υπάρξει διαχείριση μέσω της διαφοράς ενωτικά. Έτσι νομίζω ότι στο μέλλον το κυριότερο θέμα που θα τεθεί θα είναι η επικουρικότητα. Όχι μόνο με την έννοια που το λένε συνήθως, αλλά και για να επιτρέψει στον καθέναν από εμά να διατηρήσει μέσα στο κοινό, αυτό πλαίσιο, τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καμία ανθρώπινη κοινωνία μέχρι την Ένωση δεν αντιμετώπισε παρόμοια πρόκληση nous Ευχαριστώ για τη σαφήνεια αυτή. Και τώρα και τώρα λέγω αν δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο ή απορία καιρός θα ήταν να βγάλουμε τα συμπεράσματα του ενδιαφέροντος αυτού σεμιναρίου των τελευταίων δύο ημερών. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο γι' αυτό στην κυρία Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ δύσκολο καθήκον να συνοψίσει κανείς όλα όσα υπόθηκαν χθες και σήμερα εδώ. Γιατί τα θέματα είναι πολύπλοκα. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει η ορμή τώρα στη ζωή της Ένωσης για το θέμα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνθήκη της Λισαβόνας τα έχει περιλάβει στο πρωτογενές δίκαιο και στην ιδρυτική συνθήκη. Και τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλα. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον τομέα αυτόν που είναι ταυτόχρονα και μια βαριά ευθύνη. Γι' αυτό θα ήθελα να ξανατονίσω αυτό το θέμα της ευθύνης που έχουν τα θεσμικά όργανα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία, οργανισμούς και υπηρεσίες που διαθέτουμε ώστε πράγματι να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Με χαρά άκουσα την Επίτροπο να λέει σαφέστατα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή για παραβιάσεις της χάρτας. και κατά την υποβολή νομοθετικών προτάσεων και κατά την εφαρμογή τους στο επίπεδο και μεταφοράς τους στην εθνική νομοθεσία εφόσον βέβαια αφορά κοινωτικά θέματα ενωσιακά. Και ακούσαμε και τον διευθυντή της υπηρεσίας που μας είπε και αυτός ρητά ότι βλέπει τον ρόλο του ως χορήγηση πληροφοριών και επιτήρηση για την προστασία των δικαιωμάτων που όπως είπα και πριν τα συμπεριλαμβάνει η Δυτική Συνθήκη ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε μία σωστή αλλά και οριζόντια εικόνα του τι συμβαίνει στην Ένωση. Επίσης καθήκον μας είναι να μην ξεχνάμε και τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες μέλη της Ένωσης. Παραδείγματος χάρη αυτά που είπε ο κύριος Γέροπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δεσμεύσεις αυτές. Ποιες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη από διεθνή συμβάσεις. Λοιπόν, εχθές το απόγευμα συζητήσαμε, αν δεν απατώμε, το ρόλο των δικαστηρίων σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της ορμής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα συνταγματικά δικαστήρια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι Στρασβούργο. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα δύο αυτά δικαστήρια είναι ιδιαίτερα σημαντικά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, τεράστιες. Αλλά πρέπει να δούμε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που μπορεί τελικά να αποβούν φραγμός στη σωστή χρήση. Και βέβαια δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τον ρόλο του ακαδημαϊκού κόσμου, των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μη κυβερνητικών όμικρων. Διότι αυτά τα όργανα και σώματα είναι εκείνα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και την καθημερινή εφαρμογή ή μη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό βλέπω σημαντικό ρόλο και για το Κοινοβούλιο, για να μας υπενθυμίζει ότι πολύ καλά είναι όλα αυτά μεν και θετικά, αλλά, αλλά ναι, αλλά δεν μπορούμε όλα να τα βλέπουμε μόνο στο πρώτο επίπεδο εκ πρώτης απόψεως Ξέρουμε ότι σιγά σιγά θα εφαρμοστούν, αλλά αν δεν συνδεθούν όλα αυτά με την καθημερινή ζωή και ανάγκες των πολιτών και των δύο φίλων, τότε θα, θα χαθούμε. Θα Πολύ χρήσιμο λοιπόν, πολύ χρήσιμες ήταν όλες οι παρεμβάσεις που ακούσαμε για την προετοιμασία της έκθεσής μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και νομίζω ότι ακριβώς ο ρόλος του Κοινοβουλίου έγκυται στο να ακολουθεί, να παρακολουθεί, να επιτηρεί τη λειτουργία των διαφόρων άλλων οργάνων και οργανισμών Είναι λοιπόν ρόλος ελέγχου και επιτήρησης και αντίδρασης βέβαια όταν έρχεται η ώρα για τη λήψη των αποφάσεων αν έχουμε διαπιστώσει ελλείψεις δεν θα παραλείψουμε να το δηλώσουμε. Νομίζω ότι αυτά είναι όσα μπορούσε κανείς να πει ως συμπεράσματα σε τόσο λίγο χρόνο. Πρέπει όλοι και όλες να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται εδώ γιατί είναι πολύ σημαντική και αν δεν την εκμεταλλευτούμε την ορμή αυτή τότε θα παραμείνουμε στο επίπεδο των χαρτιών δεν θα υπάρξει πραγματική αλλαγή στην καθημερινή ζωή των πολιτών ενώ στόχος μας είναι όλα αυτά να φτάσουν μέχρι τον πολίτη. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής ΕΛΕΦ ευχαριστώ όλους τους ομιλητές πολύ. Καθώς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών του ακαδημαϊκού κόσμου και όλων των οργανισμών και οργάνων που συμμετέσχουν στην ακρόαση αυτή στο σεμινάριο αυτό σήμερα και χθες. Και φυσικά ευχαριστούμε και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έκαναν τον κόπο να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση αυτή. Ιδιαίτερα η κυρία Κίνγκα Γκάλ που είναι διακεκριμένη συνάδελφος και μέλος της Επιτροπής ΕΛΕΦ, εισηγήτρια δε για το θέμα της ένταξης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε και εγκαίρως. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας επιτέλους ισχύει που είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό ιδιαίτερα. Είναι κάτι πολύ καλό, πολύ καλό. Παρά την κρίση παρά την τεράστια οικονομική κρίση που απορροφά την προσοχή όλων των θεσμικών οργάνων και παρά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παρά επίσης το γεγονός ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είχε τέτοιες σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των οργάνων γνωρίζουμε και τις διαμάχες που έχουν σημειωθεί, παρόλα αυτά η συνθήκη της Λισαβόνας αφορά κυρίως τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι βήμα τεράστιας πολιτισμικής σημασίας. Βασίζεται στην ένωμη τάξη και από την αρχή της θεσμικής μας ε, εμπειρίας γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν, υπάρχουν, αν δεν υπάρχει ένας κατάλογος δικαιωμάτων, ένα Bill of Rights που λέμε. Γιατί η ευρωπαϊκή εμπειρία κατάφερε να φτάσει ως εκεί που έφτασε χωρίς να δηλώνει μέχρι τώρα σαφώς ποιες ακριβώς είναι οι αρχές της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει έλλειψη αρχών ή ελλειπής νομολογία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά υπάρχει κάποια έλλειψη αξιών, υπάρχει τελικά, κάποια. Και αυτήν πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να φωτίσουμε άπλετα το θέμα αυτό να το συζητήσουμε ειλικρινά. Καθήκον μας είναι το θέμα αυτό αρχής να το συζητήσουμε πλήρως και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα με την συνθήκη της Λισαβόνας διότι μας δίνει το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει νέες δικαιοδοσίες να αποτελεί πράγματι μέρος του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ασφαλείας και ελευθερίας. Ε, ε. Είναι επίσης πολύ σοβαρό θέμα το ότι όλες αυτές οι νέες δικαιοδοσίες τώρα θα υπόκεινται σε έλεγχο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει αυτός ο νέος διάλογος. Ο νέος διάλογος που θα οικοδομηθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Α, αυτό δεν θα είναι βέβαια εύκολο, γιατί αρκετό καιρό το συζητάμε στην Επιτροπή ΕΛΕΦ και στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά, πολύ καλά καλύτερα από, οτε, από ποτεδήποτε πριν ότι, ότι υπάρχουν πολλοί τεχνικοί φραγμοί, τεχνικά θέματα, λεπτομέρειες, πολύπλοκες, δύσκολες και πολλές πολιτικές δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν δεν πρόκειται να λυθούν από μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος και όλα αυτά είναι πολύ απαιτητικά, πάρα πολύ απαιτητικά. Αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας δεν είχε σαν στόχο ούτως ή άλλως να διευκολύνει τη ζωή του κοινοβουλίου μας αντίθετα. Θα την δυσκολέψει. Θα είναι πολύ πιο απαιτητική και αυτή και θα είναι και πολύ πιο υπόλογο το κοινοβούλιο ενώπιον των πολιτών γιατί με περισσότερες δικαιοδοσίες και εξουσίες θα υπάρχει και μεγαλύτερη ευθύνη θα είναι πιο υπόλογο στους πολίτες παρόλα αυτά όμως τελικά νομίζω ότι ότι ότι ότι, ότι πρέπει να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν πια, δεν θέλουν πια να χωρίσουν περισσότερες δικαιοδοσίες στην Ευρώπη διότι εφόσον μάλλον αυτή δεν είναι αρκετά σαφής, δεν λέει αρκετά ρητά και ισχυρά ότι ο, το κάθε βήμα πρέπει να ακολουθείται και από πρόσθετο επίπεδο εγγυήσεων, προστασίας των δικαιωμάτων τους, των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό είναι η μαγεία της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι προσθετική, προσθετική στην ε, προηγούμενη προστασία που είχε κατακτηθεί με τόσους αγώνες μέσα στα χρόνια από τους Ευρωπαίους πολίτες, από τους Ευρωπαϊκούς λαούς, από κάθε χώρα μέλος και την συνταγματική της εμπειρία. Τώρα έχουμε μια πρόσθετη φάση. Έναν καινούργιο σταθμό στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Που είναι πολύ προωθημένος για τη νέα γενιά είναι. Και με τελείως ενημερωμένο και σύγχρονο τρόπο σφαιρικά. Δεν πρόκειται λοιπόν να βλάψουμε κανένα δικαίωμα κεκτημένο από τα χρόνια και τους αιώνες από τα κράτη-μέλη. Αντίθετα θα τα εμπλουτίσουμε όλα αυτά, θα τα διευρύνουμε και θα τα εμβαθύνουμε. Και την εμπειρία και το πρότυπο προστασίας των πολιτών όπως έχει διατυπωθεί και επιβεβαιωθεί από κάθε χώρα. Μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό, όλοι μαζί. Και σωστά, δεν θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι εύκολο. Το έχουμε δει και από τις συζητήσεις μας εδώ. Ότι ορισμένα σημεία που έθιξαν οι ομιλητές το έδειξαν. Η πρόκληση λοιπόν είναι πολύ μεγάλη και ακριβώς γι' αυτό αξίζει τον κόπο να μην ξεχάσουμε, να μην χάσουμε το δρόμο γιατί το ευρωπαϊκό καινοβούλιο δεν θα σημαίνει πλέον τίποτε αν δεν αφορά η δράση του τους πολίτες, πολίτες, πολίτες. Και τα δικαιώματα, όματα, όματα και τις αξίες. Δεν έχει κανένα νόημα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία άμα δεν υπάρχει η χάρτα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και με αυτό το καταληκτικό συμπέρασμα λύεται η συνεδρίαση αλλά και το σεμινάριο. Σας κατευχαριστώ.